Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Πολύ σημαντική η σημερινή μας συνεδρίαση. Θα ακούσουμε τους δύο εισηγητές μας, τον κύριο Φερνάνδες και τον κύριο Μπούλμαν, που θα μας παρουσιάσουν το κοινό σχέδιο έκθεσης. Θα ακολουθήσει εκτενής ανταλλαγή απόψε. Καταρχήν συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Μήπως υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, εγκρίνεται. Πρακτικά. Τη συνεδρία 23 Απριλίου, 23 Φεβρουαρίου, συγγνώμη, 26 Φεβρουαρίου και Δευτέρα Μαρτίου. Σας βρίσκουν σύμφωνος. Υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά των τριών συνεδριάσεων που ανέφερα. Όχι, οπότε και αυτά εγκρίνονται. Και να δώσω τώρα το λόγο στον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, αν θέλει να πει κάτι. Ε, Σε ευχαριστώ Πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση. Γιατί Έχουμε εδώ τους ε, συγκητές του Κοινοβουλίου που θα μας παρουσιάσουν το σχέδιο της έκθεσης που έχουν συντάξει, δεδομένη θέση του ΕΚΟΦΗΝ και σήμερα θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα παρουσιάσει ε, μια φιλόδοξη άποψη και επίσης και την ε, δέσμευσή μας. Μια που πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνος και το έχουμε διάγραμμα. έχουμε αυτή την συνεδρίαση που γι' αυτό τη συγκαλέσαμε στις 8 το πρωί εδώ στο Στρασβούργο. Και λέω λοιπόν είμαστε ε, δεσμευμένοι τόσο ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το στενό πιεστικό χρονοδιάγραμμα, τόσο ώστε να ανταποκριθούμε στο πρόγραμμα Juncker ακριβώς με τις προθεσμίες που έχουν ταχθεί. Και ευχαριστούμε τους συζητητές που μπόρεσαν να κάνουν σε τόσο λίγο χρόνο ε, την εξαιρετική δουλειά τους και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες ε, για να προχωρήσουμε. Ζω. Alors pour Οπότε, για να είναι παραγωγική συζήτηση και μια και θα ζητήσετε φαντάζομαι πολύ το λόγο, να προτείνω το εξής για τη διοργάνωση των εργασιών. Θα ακούσουμε πρώτα τους συζητητές και μετά ο κάθε ομιλητής ε, να έχει δυόμιση λεπτά για το σχολιασμό, για να προλάβουν και οι συζητητές να απαντήσουν. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, να δώσω πρώτα το λόγο στον Ζωζέ Φερνάνδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά τώρα. Καλημέρα σας καταρχήν και συγχαρητήρια στον συνεισηγητή, τον κύριο Ούντο Μπούλμαν, αλλά και θερμές ευχαριστίες ε, στους υπαλλήλους μας, στους βοηθούς μας και όλους όσους, όσοι βοήθησαν ε, σε αυτό το πρώτο βήμα που είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως λέει μια κινέζικη παροιμία η αρχή είναι το εμείς του παντός ή μάλλον ε, ένας μακρύς δρόμος ξεκινά με το πρώτο βήμα και εδώ έχουμε έναν μακρύ δρόμο αλλά θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ε, έκθεση, αυτό το δρόμο και να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας γιατί θέλουμε τον Ιούνιο να επιτευχθεί συμφωνία. Θεωρούμε ότι το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, συνιστά μια ευκαιρία δεδομένη τη αρχή τη προσθετικότητα και τη συμπληρωματικότητα. και δεδομένου ότι θέλουμε να πραγματοποιήσουμε περισσότερες επενδύσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, να άρουμε νομικά εμπόδια. Δεν μπορούμε λοιπόν να χάσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνει το Ταμείο. Φυσικά έχουμε και σημαντικές προκλήσεις για τα κράτη-μέλη, για τις περιφέρειες, αλλά και για τις μεταφορές, για την έρευνα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έρευνα, για παράδειγμα, να επενδύσουμε στην έρευνα. Θέλουμε πρώτα απ' όλα ένα αξιόπιστο επενδυτικό σχέδιο ένα σχέδιο που θα στεφτεί με επιτυχία. Ένα αξιόπιστο σχέδιο. Γι' αυτό αναμφίβολα ε, λέμε ότι η εγγύηση των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να είναι ανεπιφύλακτη, ανεφόρον και αμετάκλητη. Γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη. Γιατί τα 8 δις που πρέπει να γράψουμε στον προϋπολογισμό πρέπει να τα υποστηρίξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί το Ταμείο Εγγυήσεων των 8 δισεκατομμυρίων θα αποτελέσει τη βάση της αξιοπιστίας του επενδυτικού σχεδίου. Και στη δική μας πρόταση, την πρόταση της έκθεσης για τη σύσταση αυτού του Ταμείου Εγγυήσεων, ζητούμε και μία ευελιξία. Στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ετησίως ότι οι δύο ε, αρμόδιες για τον προπολογισμό αρχές, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να συμφωνήσουν για τη σύσταση του Ταμείου. Εμείς ε, ζητούμε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα κατά τη σύσταση αυτού του Ταμείου Εγγυήσεων. Επαναλαμβάνω, η πρικοδότηση είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ και η εγγύηση των 16 δισεκατομμύριων ευρώ πρέπει να είναι αμετάκλητη και άνευ όρων. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει ενεργό μέρος στην παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσει την ομιμοποίηση του σχεδίου αυτού, χωρίς φυσικά να θέτει ένα αμφιβόλο την απαραίτητη διάκριση των εξουσιών. Είναι προφανές αυτό. Επίσης, ε, επιδιώκουμε μία αντικειμενική απόφαση δεν θέλουμε να, εμπλέκε, να εμπλέκονται πολιτικά κριτήρια στην απόφαση επιλογής των σχεδίων ή ε, σε κάποιες, στην ανέβρεση προσανατολισμών. Αυτό είναι ο στόχο, να είναι αποπολιτικοποιημένο το σχέδιο. Αλλά ζητούμε παρακολούθηση και ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Όπω σα είπα και στην αρχή, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτό που περιμένουμε είναι προτάσει προτάσεις και λύσεις, τροπολογίες. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις τροπολογίες απαιτούμε οι προτάσεις αυτές να είναι εφικτές, όχι ουτοπικές. Γιατί αν έχουμε μια πρόταση που αφισβητεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν είναι ρεαλιστική. Γιατί μια τέτοια πρόταση θα διακυβεύσει το χρονοδιάγραμμά μας και το ίδιο το επενδυτικό πλαίσιο. Το χρονοδιάγραμμα, όπως σας είπα, προβλέπει Ιούνιο του τρέχοντος έτους, μην το ξεχνούμε. Οπότε αυτή είναι η προϋπόθεση για τις τροπολογίες, να είναι ρεαλιστικές και εφικτές. Σε πολύ λίγο διάστημα α, συζητήσαμε αυτό το θέμα, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ε, για διαλαξία στη συζήτηση. Γιατί ήμασταν από την αρχή συνεργάσιμοι και διαλλακτικοί και έχουμε και αυτή τη συζήτηση γιατί επιδιώκουμε τη συνένεση. Και θα ήθελα να χαιρετήσω το έργο του συνεισηγητή Μπούλμαν. Θεωρώ ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να στεφθεί με επιτυχία αυτό το επιθυμητό από όλου επενδυτικό σχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σούντο Μπούλμαν. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καταρχάς ε, και εγώ να ευχαριστήσω, όπως και ο Ζωζέ Μανουέλ, όλους τους συνεργάτες μας που μας επέτρεψαν να επιτελέσουμε πολύ γρήγορα αυτό το καθήκον. Γιατί ήταν αναγκαίο αυτό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους συγητές, τους σκιώδεις, αλλά και τις υπηρεσίες που μας επέτρεψαν να έχουμε και τα κείμενα τόσο σύντομα τις μεταφραστικές υπηρεσίες, όλοι οι οποίοι με τη συμβουλή και την δραστηριότητά τους ε, μας βοήθησαν και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Ζωζέ Μανέλ με τον ήρεμο τρόπο με τον οποίο μας βοήθησε να καταλήξουμε στη σωστή οδό. Οι Πορτογάλοι, Ζωζέ Μανέλ, έχουν μεγάλη παράδοση στην αυσιπλοεία. Πάντα σχεδίαζαν καταπληκτικού χάρτε που επέτρεπαν να φτάσει κανεί στον προορισμό του. Έτσι πιστεύω ότι και εμεί θα το καταφέρουμε. Περί τίνο πρόκειται. Το έχουμε πει επαρκώ. Το σχέδιο αυτό επενδύσεων έπρεπε να το έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίμενε πολύ καιρό κάποια επιτροπή, τώρα έχουμε την επιτροπή Juncker, δόξα τω Θεώ, επιτέλους να μας κάνει μια πρόταση για το πώς θα μπορούσαμε ως Ευρωπαίοι να επενδύσουμε περισσότερο στο δικό μας μέλλον. Το Κοινοβούλιο, οι επιτροπές οι οποίες συναρμόδιες θα κάνουν ό,τι μπορούν ούτως ώστε ταχαίως και αποτελεσματικά να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Όμως ε, καταρχάς πρέπει να αναφερθώ σε μια απογοήτευση με την οποία πρέπει να ζήσουμε. Ελπίζω να είναι μόνο σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Τα κράτη-μέλη και λυπούμεθα γι' αυτό δεν ακολούθησαν, δεν ανταποκρίθηκαν στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις χρηματοδοτήσεις τους. Το θέλουμε αυτό για να παίξει το ρόλο του ως μόχλευση. Θα έπρεπε λοιπόν να συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη για να αυξηθεί και η δυνατότητα παρέμβασης του Ταμείου. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε, είπα τα κράτη-μέλη, αλλά η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία ανήγγυλαν ότι ναι μεν δεν θα συμμετάσχουν στο Ταμείο, αλλά μέσω εθνικών ε, ιδρυμάτων χρηματοδότησης ή μέσω συγχρηματοδοτήσεων θα συμβάλλουν. Ε, χαιρετίζουμε αυτό το γεγονό και καλούμε και τα άλλα κράτη-μέλη να, επαναλάβουν, να μιμηθούν το παράδειγμα. Αυτό τι μας λέει. Ότι η συνεργασία μεταξύ του ΕΦΣΥ και των επιτόπου φορέων των εθνικών επενδυτικών ιδρυμάτων, των περιφερειακών ιδρυμάτων, των ιδιωτικών επενδυτών, αυτή η συνεργασία όλων αυτών είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό θέλω να πω στους συναδέλφους της Επιτροπής ε, Οικονομικών. Πρέπει να προσέξουμε να λειτουργεί σωστά αυτή η συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πρέπει να τίθεται θέμα just retour. Δεν θέλουμε να υπάρξει επανεθνικοποίηση του προγράμματος αυτού. Τα κριτήρια πρέπει να είναι ευρωπαϊκά. Παρόλα, ευρωπαϊκά. Παρόλα αυτά, πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες ούτως ώστε να υπάρξει η καλύτερη συνεργασία για να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, να συμμετέχουν οι περιφέρειες στις εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Επ' αυτού πρέπει να εργαστούμε, να βρούμε ευφυείς λύσεις. Και θα κάνουμε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θέλουμε η Επιτροπή Επενδύσεων που προβλέπεται που θα μελετάει κατά πόσο είναι αξιόπιστα τα προγράμματα και κατά πόσο είναι αρκετά όρημα για να μπορέσουν να ε, αποσταλούν με κατόπιν για ε, έγκριση από τις ε, ευρωπαϊκές αρχές. Θέλουμε λοιπόν σωστές επενδύσεις. Συμφωνώ με τον Ζωζέ Μανέλ. Δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τίποτα που ήδη χρηματοδοτείται. Δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε αφαιρώντας από αλλού χρηματοδότηση. Θέλουμε να υπάρχει συμπληρωματικότητα και πρέπει να την ορίσουμε αυτήν την προσθετικότητα καλύτερα ας πούμε. Πρέπει να είναι οι πιο ε, ρηψοκίνδυνες επενδύσεις που μέχρι στιγμής δεν χρηματοδοτούνται και που θα μα βοηθήσουν να καλύψουμε κενά στην ευζωνικότητα, στις μεταφορές, στη βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον εξυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής μας και για τις επενδύσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα. Γι' αυτό δεν θα σας εκπλήξω ότι το άρθρο 5.2α καθορίζονται επενδυτικά κριτήρια που μιλάνε για περισσότερο κίνδυνο, για προσθετικότητα και για συνολική οικονομική αποδοτικότητα. Τρίτο σημείο. Πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το ταμείο. Φυσικά θα βασιστούμε πολύ στην τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και στο άρθρο 4 λέμε ότι πρέπει να υπάρχει η εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούν να κινητοποιηθούν τα αναγκαία ποσά. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα χορηγεί την εγγύηση. Οπότε θα πρέπει να φέρει και τον κίνδυνο. Είτε μέσω του first loss, είτε γενικότερα ως εγγύηση. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφές ότι ο κίνδυνος θα φέρετε αποκλειστικά από τον ενωσιακό προπολογισμό. Λοιπόν, κοιτάξτε, ας κάνουμε ένα πείραμα. Στο τέλος ε, της συνεδρίασης δώστε μου τα πορτοφόλια σας, δώστε μου τις πιστοτικές κάρτες, δώστε μου αποσπάσματα του λογαριασμού σας και θα τα επενδύσουμε. Ο Ζωζέ Μανέλ και εγώ τι θα πείτε. Θα πείτε ναι φίλε, σας πιστεύουμε, είστε πολύ συμπαθείς, ε, ποτέ δεν μας έχετε εξαπατήσει. Αλλά ποιος θα είναι ο διαχειριστής των επενδύσεων, ποιος θα ελέγχει ότι είναι λογικές επενδύσεις. Σας πιστεύουμε, αλλά πρέπει να βλέπουμε σε ποιο χαρτοφυλάκιο θα επενδύσετε. Γιατί είναι δικά μας τα λεφτά που σας δίνουμε. Η ίδια κατάσταση ισχύει και γενικότερα. Και δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια τέτοια κατάσταση θα πει ναι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λειτουργήσουν αυτές οι εγγυήσεις αλλά έναντι των ψηφοφόρων έναντι των φορολογουμένων μας. Θέλουμε κάποιες ε, διαβεβαιώσεις ότι όλα αυτά θα πάνε καλά όπως ε, μας παρουσιάζεται. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν πρόκειται για υπερβολική γραφειοκρατία. Δεν πρόκειται για υπερβολική επιφλακτικότητα Είναι ουσιώδης πολιτική λόγη Γι' αυτό λέμε θέλουμε να υπάρχει δημοκρατική λογοδοσία. Θέλουμε να υπάρχει ένα σύστημα όπου θα ενημερωνόμεθα αλλά θέλουμε να έχουμε και το λόγο μας όταν ε, θα γίνουν για παράδειγμα θα ληφθούν οι αποφάσεις για τις ηγετικέ θέσεις αυτού του οργανισμού και για το ποιοι θα αποφασίζουν όχι να υποκαταστήσουμε άλλα θεσμικά όργανα θέλουμε να βοηθήσουμε να υπάρξουν καλές προτάσεις δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό νομίζω ότι είναι απλώς η υποχρέωσή μας ευχαριστώ πάρα πολύ Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα. Όποιος θέλει έξι μόνο μπορεί να λάβει το λόγο. το Με το λέει, σχετικά με αυτά που είχαμε από τους ε, συνεισηγητές, φερναντές και Μπούλμα. Κύριε Γκάρδια Θάβολ, πρώτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να προσθέσω και πάρα πολλά, μια που ήδη μας μίλησαν δύο συνεισηγητές, αλλά τέλος πάντων ε, έχουμε συνεργαστεί ε, στενά με τους συνεισηγητές αυτούς εδώ και μπορέσαμε να δούμε ακριβώς τι προτείνουν ε, εμείς από πλευράς προϋπολογισμού, από πλευράς ομάδα ομάδας και τις βασικές μας προτάσεις τις έχουν καλύψει στο σχέδιο κειμένου που και οι δυο τους συνέταξαν. Ο Χωσιμονών μας μίλησε πριν για ευελιξία, μα στον προπολογισμό είναι κάτι το οποίο το επικαλούμε στα συνέχεια. Από την αρχή είπαμε ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και όταν έγινε ε, η η διαπραγμάτευση για το δημοσιονομικό πλαίσιο είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε την ευελιξία για να μπορεί σε κάποιες εξωτικές περιστάσεις να προσαρμοστεί ο προπολογισμό. Για ακριβώ δεν ξέραμε ότι θα υπάρξει το πρόγραμμα, το σχέδιο Juncker. Και γι' αυτό λέμε τώρα ότι ό,τι μπορούμε από πλευρά ευελιξία να το επιστρατεύσουμε για να γίνει σχετική προοικοδότηση. Έχουμε τώρα αυτές τις προτάσεις να τις ε, συζητήσουμε. είπαμε να, να αποφασίσουμε σήμερα το Connecting Europe Facility, το Horizon 2020, ε, όλα αυτά τα οποία έχουν κοστίσει αρκετά. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε ό,τι θα χρειαστεί στο μέλλον, να μπορέσουμε να προοικοδοτήσουμε αυτό το εγκυβδοτικό ταμείο ε, και λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε περικοπές από τα προγράμματα αυτά που προανέφερα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν χρειάζεται, γιατί με την παρούσα πρόταση η εγγύηση που χρειάζεται για το πρόγραμμα Juncker ε, δεν βρίσκεται εν κινδύνο. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να το στείλουμε ξεκάθαρο. Επίσης πολλές από αυτές τις προτάσεις κατατείνουν στο ότι τα 16 αυτά δις υπάρχουν στον προπολισμό και ό,τι και να γίνει θα υπάρχει αυτή η εγγύηση. Πάντως ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει κατά τη χρήση του 2017 και για διαφορετικούς ε, λόγους είπαμε ότι το πρόγραμμα δεν θα εκτελεστεί όπως είχαμε προβλέψει το 2015. Έχουμε 490 εκατομμύρια από το ΙΤΕΛ γιατί δεν προχώρησε το πρόγραμμα ακριβώς όπως ε, περιμέναμε και είπαμε προτάθηκε αν χρειαστεί να κόψουμε κάποια, ε, κάποιους πόρους από το Connecting Euro Facility από το Horizon 2020 και από την κατηγορία 1α για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το σχέδιο Juncker. Επομένω, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι νυφαλιότητα. Γιατί η πρόταση στέκει πάρα πολύ καλά και από τεχνοκρατικής απόψεως είναι άψογη και επίσης δεν ε, θίγουμε καθόλου το Ταμείο Εγγύσεων και μπορεί αυτό να λειτουργήσει με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τάβης Επενδύσεων. Το Συμβούλιο επίσης έχει 1,5 χρόνο, εν συγγνώμη 1,5 μήνα για να ε, λάβει υπόψη, να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με αυτό το οποίο προτείνουμε. Και ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Όντως πρέπει να πείσουμε το Συμβούλιο. Ο κύριος Νούνες. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, κυρία Άσχορτ, δυστυχώ απουσιάζει. Πάντω, ε, μίλησε εκτενώ μαζί του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών για να αποκρισταλώσουμε τη θέση τη ομάδα μα του ECR. Το επενδυτικό χάσμα στην Ευρώπη είναι κυρίω αποτέλεσμα τη έλλειψη ανταγωνιστικότητα. Οπότε θα προσπαθήσω στα δυόμιση λεπτά που μου δώσατε να περιοριστώ σε ορισμένα σημεία. Μια και αντιμετωπίζουμε όμως αυτή την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα του ΕΦΣΙ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, δεν θα πρέπει να είναι εναλλακτική λύση το υποκατάστατο των υγιών οικονομικών ε, ή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Βέβαια, ε, αναγνωρίζουμε ότι είναι έκτακτη η κατάσταση, έκτακτη καιρή και άρα θα πρέπει να λάβουμε και έκτακτα μέτρα που κατά τη γνώμη μας όμως θα πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Γι' αυτό έχει νόημα να μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και κάποιες προσπάθειες που θα αναλάβουμε σε επενδυτικό επίπεδο, αλλά θα είναι περίεργο να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, σημερινή επενδυτική κατάσταση στην Ευρώπη. Ε, οπότε θα πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα τα κονδύλια του ΕΦΣΥ. Και όχι ΕΦΣΥ, μάλλον ΕΞΥ, δηλαδή ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο ή Ευρωπαϊκή Εγγύηση Στρατηγικών Επενδύσεων και όχι Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θέλουμε φυσικά τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στο Ταμείο και φυσικά να γίνεται ανεξάρτητη και αξιοκρατική επιλογή των σχεδίων ανάλογα με την οικονομική βιωσιμότητά τους, ώστε γιατί αν δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια τα κράτη-μέλη δεν θα ενθαρρυνθούν για να συμμετέχουν στο Ταμείο με συνεισφορές. Δεν μας αρέσουν τα κριτήρια της γεωγραφικής κατανομής ή ο ρόλος ε, της Επιτροπής Επενδύσεων ε, ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα δικαιώματα ψηφοφορίας που θα έχουν τα κράτη-μέλη που θα συνεισφέρουν στο Ταμείο. Ίσως το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι το Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θα πρέπει να υπονομεύει τι συμφωνίε για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί μιλάμε για ένα ταμείο που εντάσσεται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αλλά είναι σημαντικά τα θέματα τη βασική, τη θεμελιώδου έρευνα. Δεν θα πρέπει να υπονομευθεί από μεταφορά των κονδυλίων στο ταμείο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μούρεσαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω δύο-τρία σημεία τα οποία θα ήθελα να σας αναφέρω. Πρώτα πρώτα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι την υποχρέωση λογοδεσία αλλά και την διαφάνεια στα πλαίσια του Ταμείου Στατικών Απαντήσεων, ώστε να λειτουργήσει όπω πρέπει. Οπότε και θα πρέπει και εγώ να σας τονίσω ότι οποιαδήποτε ανάμειξη τη πολιτική και των πολιτικών όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και έργων, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αλλά βέβαια θα πρέπει να βρούμε τα επαρκή μέσα, ώστε να γίνεται δημοκρατικό έλεγχο και κυρίω να μην υπάρχει δυσλειτουργία αυτών των δεσμικών οργάνων τα οποία θα έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση του Ταμείου Στατικών Επενδύσεων. Οπότε γι' αυτό και σα λέω ότι είμαι κατά ορισμού της Επιτροπής Επενδύσεων από τους ε, πολιτικούς. Οπότε θα πρέπει και εμείς να ασκούμε έλεγχο και να υπάρξει κάποιο σύστημα να περνούμε από ακρόαση τους ε, υποψηφίους αλλά θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος για το Διευθυντικό Συμβούλιο και οι διορισμοί να γίνονται επί τη βάση των ε, ικανοτήτων και δεξιότητων. Τώρα, όσον αφορά το Ταμείο Εγγύσεων νομίζω θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία, όπως λέει και η έκθεση του Κοινοβουλίου, ακριβώς όπως είπαν και οι Να δούμε τι θα γίνεται κάθε χρονιά, ούτως ώστε να μην υπάρχουν φραγμοί στην ε, εκτέλεση των προγραμμάτων, θα πρέπει και αυτά τα 80 δις να είναι διαθέσιμα, με, τα 8 δις να είναι διαθέσιμα και ε, επίσης οι χρηματαγορές να αποδίδουν αξιοπιστία σε αυτό το ταμείο, σε αυτό το κεφάλαιο 8 δις. Είπε ο κύριος Μπούλμαν επίσης κάποια πράγματα σχετικά με την ε, συμμετοχή των κρατών μελών. Σε αυτή τη φάση ακόμα δεν έχουν συμμετάσχει, αλλά νομίζω ότι αυτό ε, ισχύει γιατί ακόμα δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα ώστε τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν. Δηλαδή, ε, πώς θα συμμετάσχουν, πώς θα ψηφίζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, νομίζω ότι επομένω είναι ανεπαρκή ακόμα αυτά τα κίνητρα και αν θέλουμε να ελκύσουμε τα κάτι μέλη στο μέλλον θα πρέπει ακριβώ να επεξεργαστούμε κάποια άλλα κίνητρα και να τους ελκύσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για το πολύ αξιόλογο έργο τους και να συμφωνήσω με τα συγχαρητήρια και προς τους σκιώδεις εισηγητές. Σε τελική ανάλυση δεν θέλουμε μια πολιτικοποιημένη διαδικασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια στο σχεδιασμό και μια ασφάλεια δικαίου. Το μέχρι τώρα έργο ήταν εξαιρετικό. Αλλά φυσικά επιδέχεται κάποιες βελτιώσεις. Αυτό που ε, είπα ισχύει για την Επιτροπή Επενδύσεων και για το πώς θα γίνεται η επιλογή των προγραμμάτων. Ε, αν υπάρχει ένας πολύ μακρύς κατάλογος σωρευτικών υποχρεώσεων και προϋποθέσεων ε, δεν θα είναι θετικός. Πρέπει να εστιάσουμε στην ποιότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των προγραμμάτων. Επιπλέον, θεωρώ ότι είναι ουσιώδες να μην δημιουργήσουμε νέα γραφειοκρατικά εμπόδια μέσω της λειτουργίας αυτού του Ταμείου. Βεβαίως αυτά που λέγονται έχουν ε, κάθε αιτιολόγηση αλλά πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και το ΕΦΣΙ και η Τράπεζα Επενδύσεων και αν πρέπει να περάσουν και από διάφορες περιφερειακές και τοπικές αρχές θα έχουμε επιπλέον γραφειοκρατικά εμπόδια. Διαρωτώ με λοιπόν. Ε, και τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αυτή η επιπλέον γραφειοκρατία στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ούτως ώστε να είναι κάτι σωστό. Εάν έχει έννοια ένα πρόγραμμα και επ' αυτού πρέπει να επικεντρωνόμεθα, αυτόματα θα έχει θετικό αποτέλεσμα στην απασχόληση. Πρέπει να εκφράσω τον σκεπτικισμό μου για το λεγόμενο αυτό κόμβο ε, διαβουλέψεων. Το κόμβο επενδυτικών συμβούλων. Δεν ξέρω εάν έχει έννοια να έχουν τόσα καθήκοντα ε, αν θα έχει κόστος ε, ή όχι δεν το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε μέσω μιας επιπλέον επιλογής για το ποιος θα, ε, ποια προγράμματα θα περνάνε από αυτό το κόμβο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα και όχι μεγάλος αριθμός προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζάνι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οπωσδήποτε η πρόταση των δύο συνεισηγητών είναι ένα μικρό βήμα προς την σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπωσδήποτε είναι κάτι το θετικό γιατί εστιάζεται περισσότερο όσον αφορά τον χαρακτήρα αυτών των έργων, όσον αφορά ε, την προσθετικότητα, όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου και επίσης τις ε, μη πράγματα τα οποία ε, δεν είχαν περιληφθεί με αυτόν τον τρόπο στην αρχική πρόταση. Επομένως, πρόκειται για βήμα πρόοδο όσον αφορά την διακυβέρνηση και περισσότερη υποχρέωση λογοδοσίας. Παντός χρειάζεται ακόμα περισσότερη διαφάνεια, κυρίως όσον αφορά την λειτουργία σε κάθε επίπεδο όσον αφορά το Ταμείο. Οπότε, ε, όσον αφορά αυτό τον κόμβο συμβουλών, υπάρχει ε, μια δυσπιστία, σκεπτικισμό για αυτά τα 10 εκατομμύρια για να δούμε πώ θα προχωρήσει. Ε, για να δούμε τώρα κάποια άλλα σημεία. Δεν είναι ακόμα τα πράγματα τόσο σαφή όσον αφορά τα κριτήρια των επενδύσεων. Άρα αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει. Όσον αφορά τώρα τους πόρους, κατά τη γνώμη μου, Με αυτή την προσέγγιση θα καλυφθεί η γενική ανάγκη και θα υπάρχει ευελιξία. Όμως, προσοχή, γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά τον ισολογισμό και όσον αφορά τους επενδυτές. Άρα χρειάζεται να γίνει επανεξισορρόπηση του προϋπολογισμού για να δούμε τι θα γίνει με τους πόρους που θα πάνε στις υποδομές και από την άλλη μεριά τους πόρους για τις ΜΜΕ. Θα πρέπει να λυθούν περισσότερο υπόψη ΜΜΕ γιατί εκείνες είναι το μηχανή της οικονομικής πρόοδου. Άρα να δούμε πώς θα ωφεληθούν περισσότερο εκείνα τα προγράμματα και έργα που φέρνουν ε, περισσότερη ωφέλεια οικονομική ή και από πλευράς περιβάλλοντος και μακροπρόθεσμο. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την ιδιωτικοποίηση των κερδών. Και οπότε αυτό το trade να προσπαθήσουμε να το ρυθμίσουμε καλύτερα. Ο κύριος Μπέγκε, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι για μένα η χρηματοδότηση αυτού του νέου μηχανισμού. Ναι στα προγράμματα, και με βάση την πείρα που έχουμε από τις ε, κοινέ ε, επιχειρήσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το PPP. Έχει έρθει ο χρόνος για τέτοιου τύπου προσπάθειες αλλά το πόσο καλά θα πάει θα το δούμε κατά την εκτέλεση του επόμενου προπολογισμού γιατί το θέμα της αξιοπιστίας και της δυνατότητας των θεσμικών οργάνων να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο θέμα και να το αποφασίσουν σύντομα και αποτελεσματικά, όλα αυτά μας ενδιαφέρουν όλους. Μιλήσαμε επίσης για προγραμματισμό και για κράτος δικαίου. Οπωσδήποτε, βεβαίως, πρέπει να ισχύει, όπως για όλα τα εγχειρήματά μας. Πρέπει όμως επιτέλους η Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία ούτω ώστε να έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο για το πώς θα εκτελούμε τα προγράμματα. Θέλουμε να χρονοτριβούμε τόσο πολύ όπως ε, κάνουν κράτη-μέλη για να χτίσουν μια γέφυρα και βεβαίως δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να μειωθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα κανενός αλλά δεν είναι δυνατόν να αλληλοτροχοπεδούμεθα στις προσπάθειές μας για να υπάρξει ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Μία παρατήρηση για την πρόταση της Επιτροπής. Μου είπαν σε συζητήσεις ότι πήραμε την απλούστερη λύση για τη χρηματοδότηση, αλλά η απλούστερη δεν είναι πάντα πιο αποτελεσματική. Και δεν νομίζω ότι προσβάλλω κανέναν ε, στην Επιτροπή όταν λέω ότι πρέπει να δούμε και τι εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν. Θα μπορούσε να διευκρινίσει καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα, είχαμε τα συγκυριακά προγράμματα Μπαρόζο 1 και 2 στο παρελθόν, και είχαμε και το μέσο για τα τρόφιμα το 2008 τότε είχε υπάρξει δημιουργικότητα και ετοιμότητα να επιτύχουμε πράγματα που τώρα ε, αποκλείονται εκ των προτέρων. Και επίσης το θέμα της έρευνας. Έχουμε αποτελέσματα ναι. μετά από ε, μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για το πολιετές πρόγραμμα για την έρευνα και δεν είναι δυνατόν τώρα να αφισβητούνται Και για την ε, διαγραφή των 18 και 19 ως βάση χρηματοδότησης νομίζω ότι είναι καλή αρχή. Πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικά για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τις εγγύησεις και όχι ευθύς εξ αρχής να κάνουμε τέτοιες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκια. Ευχαριστώ. με ανησυχεί πόσο επιμένουμε στην ε, πίεση χρόνου για να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί σύντομα το ΕΦΣΥ. Γιατί η πίεση του χρόνου δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Ιδίω ε, για τόσο σημαντικά εγχειρήματα που θα πρέπει να οδηγήσει σε επενδύσεις 300 δις. Αν τα έχουμε αυτά τα χρήματα δεν χρειαζόμασταν ευσύ τους ή Να αναφέρω δύο θέματα που νομίζω ότι πρέπει να σε απασχολήσουν περισσότερο από ό,τι μέχρι τούδε. Το πρώτο είναι ότι το ΕΦΣΙ θα δώσει κρατικές επιδοτήσεις. Είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται. Πρέπει να έχουμε υπόψη ποιες είναι οι συνθήκες για να δίνονται τις επιδοτήσεις. Ε, δεν αναφέρονται αρκετά στο κείμενο επ' αυτού. Οπότε πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι συνθήκες της αγοράς όταν χρηματοδοτούμε προγράμματα. Διότι το μεγαλύτερο τμήμα των χρηματοδοτήσεων θα είναι ιδιωτικέ επενδύσεις. Άρα πρέπει να υπάρχουν κέρδη για να επενδυθούν. Τα κέρδη τα αποκομίζει κανείς μετά από ανταγωνισμό με άλλους. Ενώ οι ε, επιδοτήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Είτε δεν υπάρχει, ε, είτε δεν, υπάρχει, δεν συμμετέχουν αυτές οι επιδοτήσεις σε τομείς της αγοράς όπου υπάρχει ανταγωνισμός, οπότε ενισχύουν μονοπωλιακές καταστάσεις. Πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά. Δεύτερον, απαιτείται λέγεται προσθετικότητα. Ο κύριος Μπούλμαν είπε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την προσθετικότητα μέσω προγραμμάτων που είναι πιο ρηψοκίνδυνα από αυτά που συνήθως χρηματοδοτεί η αγορά νομίζω ότι είναι απατηλή αυτή απατηλό αυτό το συμπέρασμα ο υψηλός κίνδυνος μπορεί να επιδιώκεται περισσότερο ή να χαρακτηρίζεται ως υψηλότερος για να λάβει κανείς χρηματοδότηση προγράμματα δηλαδή που ούτως ή άλλως θα χρηματοδοτούνται να χρηματοδοτούν από αυτό δεν χρειάζεται λοιπόν να επιδιώξει κανείς από την άλλη να είναι πιο ρηψοκίνδυνο το πρόγραμμά του για να είναι σίγουρος ότι θα λάβει χρηματοδότηση. Οπότε δεν βλέπω να εγγυόμεθα την προστατικότητα. Ευχαριστώ κύριος Ντονανό. Κύριε Πρόεδρε, σίγουρα χρειάστηκε πολλής χρόνος για να καταλάβουμε ποιες ήταν οι βασικές, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου. Κατάλαβα, κατάλαβα ότι πρόκειται τελικά για ένα σύστημα εγγύσεων. Εμεί ελπίζαμε ότι θα είναι ένα θέμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά τελικά είναι ένα πρωτότυπο σχέδιο που θα στηρίζεται σε τραπεζικέ επενδύσει. Εντάξει. Ο κύριο Φερνάνδες μίλησε για μια στη βαρότητα της εγγύησης, θα πρέπει να είναι αμετάκλητη και σταθερή. Αυτό όμω δεν αποκλείει την ευελιξία τη εγγύηση. Και ευχαριστώ τον εισηγητή που ακολούθησε αυτή την κατεύθυνση της ευελιξίας. Θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι όμως με αυτό το θέμα, γιατί θα ήταν κρίμα να στερηθούμε χρηματοδότησης, ε, ιδιαίτερα για την έρευνα, περιορίζοντας την ευελιξία. Και εκεί ελοχεύει ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος, γιατί η βασική και η εφαρμοσμένη έρευνα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γιουνκέρ μας είπε ότι δεν μπορούμε να ξοδέψουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ε, εννοείται. Είναι αυτονόητο. Ε, κανένας όμως δεν μας εμποδίζει να αναζητήσουμε χρήματα. Και εκεί είναι που έχουμε κενά. Γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να βρούμε κοινοτικού πόρους, όπως το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μόνο μία χώρα άρχισε να σκέφτεται αυτό το θέμα σοβαρά. Γιατί να μην έχουμε ε, ένα κοινωνικό φόρο ή ένα φόρο διοξιδίου του άνθρακα στα σύνορα. Υπάρχουν δυνατότητες ε, φορολογικών εσόδων ή η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Γιατί να μην επιβάλλονται πρόστιμα, ε, αδρά πρόστιμα για φορολογικές απάτες. Έτσι θα βρούμε κονδύλια και για να ενισχύσουμε τις εγγύησεις, αλλά και να είμαστε πιο φιλόδοξοι στα επενδυτικά μας σχέδια. Τώρα, στο θέμα των εγγύησεων, έχουμε και τις εθνικές τράπεζες και τις περιφερειακές ίσως που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στις εγγύησεις. Γιατί όχι, γιατί να μην αναμίξουμε και τις τράπεζες στο μηχανισμό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα προτιμούσα να μην ε, ε, θίξουμε την ε, βασική έρευνα ή την Ενεργειακή Ένωση, γιατί μιλούμε πολύ για ενέργεια, για ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασύνδεση, αλλά δεν μιλούμε για την έρευνα σε ενεργειακά θέματα, κακώς, γιατί εκεί υπάρχει πραγματικά τεράστιο δυναμικό ε, και στο πυρηνικό υδρογόνο και στο ε, μοριακό υπάρχουν πολλές δυνατότητες να βρούμε κονδύλια από την έρευνα. Ευχαριστώ κύριο Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα για τον προϋπολογισμό και δεύτερον για την επιλογή των προγραμμάτων εάν μου Πρώτα πρώτα θέλω να σας πω ότι άκουσα την παρουσίαση που έγινε στην αρχή για το σχέδιο Γιούνκερ και εντύπωσή μου είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινωνικού προπολογισμού και το Συμβούλιο. Καταρχήν δεν είχε πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε όμως ότι έχει πρόβλημα το Κοινοβούλιο. Πώς θα εμπλακεί επομένω σε αυτή την υπόθεση ο κοινωνικός προπολογισμό σαν παράγος εγγύσεων. Οπότε βλέπουμε τελείως διαφορετική μεθοδολογία τώρα όσον αφορά την εγγυητική κάλυψη. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Δηλαδή να πάμε πάνω από την οροφή που προβλέπεται από το δημοσιονομικό πλαίσιο και το Συμβούλιο. Έτσι ήθελε να κάνει. Αλλά δεν ξέρω αν το προσπαθήσαμε όσο έπρεπε. Το Κοινοβούλιο θέλει να κινηθεί κάτω από αυτά τα τόσο, αυτούς τόσο, τόσο αυστηρές οροφές, τα όρια και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται το ότι έχουμε 14% 9 στους 10 που ζητούν να συμμετάσχουν σε ελληνικά προγράμματα απορρίπτονται. Τώρα στις ε, τροπολογίες είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια δύση αναθεώρηση. Αυτό είναι καλή πρόκληση για το Συμβούλιο και Όντως έτσι έχει περισσότερη αρμοδιότητα ελεγκτική το κοινοβούλιο. Όμως έτσι αυξάνουμε την αβεβαιότητα και δυναμητίζουμε το σχέδιο Γιούγκερ. Επίσης, όσον αφορά αυτό το αποθεματικό επιδόσεων, χρειάζεται ομοφωνία πλευρά Συμβουλίου. Και νομίζω ότι αυτό δύσκολα θα επιτευχθεί. Γιατί μιλάμε για στη συνοχή, μιλάμε για αυτέ τι σκληρές διαπραγματεύσει του ενός της. Άρα χρειάζεται να είμαστε δημιουργικοί όσον αφορά αυτά τα σκληρά αριθμητικά στοιχεία στην αρχή της διαδρομής. Καλά για τη συνέχεια των επαναδέσεων, αλλά στην αρχή θα πρέπει να είμαστε κάπως προκλητικοί προς το Συμβούλιο. Προτάσουμε, δεν έχουμε χρόνο να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από αυτή την πολιτικοποιημένη λίστα των προγραμμάτων, πώς θα προχωρήσουμε στο θέμα της επιλογής, γιατί και εδώ πέρα υπάρχει ένα μυστήριο που πλανάται. Ευχαριστώ κύριο Σέκουτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές για την έκθεσή τους που βελτιώνει θεωρούμε την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θεωρούμε ότι είναι καλή έκθεση. Ως πράσινη, θα εστιάσουμε σε τρία κυρίως θέματα που είναι κέντρα βάρους και της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα είναι η διακυβέρνηση, Ακούω ότι κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιήσουμε την επιλογή των προγραμμάτων. Συμφωνώ. Αλλά να λάβουμε υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να δαπανηθούν σωστά. Γιατί αφαιρεί χρηματοδοτήσεις από τον ενωσιακό προϋπολογισμό για τον οποίο είμαστε συνυπεύθυνοι. Άρα οι εγγυήσει και πληρωμές αυτές πρέπει να έχουν σκόπιμα αποτελέσματα. Καλό είναι λοιπόν που θέλουν οι συγκητές να ενισχυθεί η ε, δομή διακυβέρνησης. Τώρα το από πού έρχονται τα χρήματα αυτά, αυτό θα αφήσω το συνάλφο έρνες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Εγώ θα ασχοληθώ κυρίως με τα κριτήρια. Ναι, βλέπω κάποιες βελτιώσεις, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά κενά πολλές δυνατότητες διαφυγής αν δούμε πώς έχουν περιγραφεί τα κριτήρια. Το πιο βασικό είναι οι επενδύσεις μας μέσω αυτού του προγράμματος να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στους στόχους του 2020 και τους μακροοικονομικούς, για παράδειγμα, να έχουν επίδραση στις θέσεις εργασίας και το ΑΕΠ. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε σαν να είναι η συνήθις διαδικασία. Και γι' αυτό είμαι κάπως επικριτικός έναντι της Κομισιόν που λέει μην υποβάλλετε πολλέ προτάσει για κριτήρια, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά τι λέει αυτό το Ταμείο. Στρατηγικέ επενδύσει Δεν είναι η συνήθι διαδικασία. Άρα δεν πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ω τη συνήθι διαδικασία. Ερώτηση προ την Κομισιόν. Στο άρθρο 1 έχουν ένα νέο ορισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να έχουν 3.000. Ενώ ο συνήθις ορισμός για τις μικρομεσαίες είναι 250 εργαζόμενες. Οπότε αυτό δημιουργεί τεράστια σάφεια για τα κριτήρια του 5, στο άρθρο 5, όπου αναφέρονται πολλά κριτήρια, συν σε ποιε μικρομεσαίε θα πάει. Αλλά αν είναι τόσο μεγάλε οι μικρομεσαίε, τότε όλοι θα μπορούσαν να πάρουν αυτέ τι χρηματοδοτήσει. Υπενθυμίζω, μικρομεσαίος μέχρι τα, τους 250 εργαζόμενους είναι ήδη 67% της απασχόλησης στην Ευρώπη. Είναι ήδη λοιπόν τεράστιο ποσοστό. Γιατί λοιπόν διευρύνεται τόσο πολύ ο ορισμό των μικρομεσαίων. Πρέπει να καλύψουμε αυτήν την ε, λαθασμένη διατύπωση. Ευχαριστώ κύριο Στόρβαλτς. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους συνεισηγητές Φερνάντες και Μπούλμαν. Πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε κάποια προβλήματα. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βρει την εύκολη λύση. Αλλά αυτό θα μας ε, κάνει ευάλωτους στους εκβιασμούς. Γιατί αν δεν πάμε με το μέρος τους, ε, ε, εκείνοι θα θυμώσουν και εμείς πρέπει να φοβηθούμε. Δεύτερον, πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα. Τρίτο πρόβλημα, έλλειψη ευρηματικής και δημιουργικής σκέψης. Το ανέφερε και κάποιος προλαλής σας. Αυτό που με ενοχλεί όμως περισσότερο είναι ο σχετικά πρωτόγονος τρόπος ε, που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίζει τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα ε, πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο. Θα μπορούσαν να τρέξουν στο Jacob Φούγκα και να δουν ότι οι εγγύησεις ε, αρκούν σε ένα τραπεζικό κόσμο. Αλλά αυτό γινόταν στο 16ο αιώνα δεν είναι και πολύ καινοτόμα προσέγγιση στα τραπεζικά θέματα. Τα έχουμε ξανακούσει και πολύ παλιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση εγγυήσεων προς την Ουκρανία. Αυτή δεν είναι και πολύ ε, καλή επένδυση από οικονομική άποψη. Αλλά αυτό μένει στον προϋπολογισμό και αρκούν οι εγγυήσεις. Αλλά πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτές τις προτάσεις. Είναι κάπως ε, γενικές. Επίσης, τι κονδύλια θα μεταφερθούν ε, ή πώς θα κινητοποιήσουμε. Έχουμε την, τους ίδιους πόρους, την, ε, την, την πρόταση για τους ίδιους πόρους, τα άνωτα όρια στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κύριος Μπούλμαν είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο Ευρωπαίοι. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να το αποδείξουμε αυτό. Πρέπει να τρέξω στην Ολομέλεια γιατί έχω μια παρέμβαση για το λαβράκι. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρώσω εδώ. Ευχαριστώ κύριο Σουμαραγκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει τώρα να τοποθετηθούμε σε αυτή την κοινή συνεδρία όσον αφορά τις βασικούς κανόνες για τη βιωσιμότητα και για τη λειτουργία του Ταμείου. Και οι άλλες ε, επιτροπές θα, θα ορίσουν το πεδίο εφαρμογή και θέματα πιο πολύ τομιακά. Τέλο πάντων, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής, οι προϋποθέσεις, ε, το, πώς θα λειτουργήσει το Δικό Συμβούλιο όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων. Θα πρέπει επομένω να δούμε τι λεπτομέρειε. Δεν μπορώ να είμαι εξαντλητικό τώρα, αλλά θέλω τρία θέματα να καλυφθούν ε, από την ρύθμιση και όχι μόνο σαν γενικά κριτήρια στο τελικό κείμενο. Πρώτα πρώτα, μιλούμε για έργα υψηλού κινδύνου και προσθετικότητα. Ε, μιλούμε τώρα για κοινή ανάληψη κινδύνου. Δεν υπάρχει μηδενικός ε, κίνδυνος. αυτό δεν θα ήταν ε, σωστό. Και όπως είπαμε προηγουμένως, θέλουμε να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αυτών των έργων και προγραμμάτων για μια ανοιχτή αγορά. και μην ολιγηθούμε σε ολιγοπόλια ή μονοπόλια, όπως γίνεται πολλές φορές στις οικονομίες μας. Επίσης θα πρέπει να λιάνουμε τις περιφερειακές ανισότητες. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Μείωση των ανισοτήτων δεν θα πρέπει να το δούμε απλουστευτικά το ζήτημα. Δηλαδή ότι χωρίς προϋποθέσεις ε, ε, χωρίς προϋποθέσεις θα έχουμε τους ιδιώτες να επενδύσουν και όταν βάλουμε επενδύσεις δεν θα έρθει κανείς ιδιώτης. Και είναι πάρα πολύ σωστό το ότι οι συνεισηγητές καθόρισαν με αυτόν τον τρόπο πώς θα γίνουν οι συνεισφορές. Και όπως είπαν, να έχουμε την αναγκαία ευελιξία. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποια περιθώρια, τουλάχιστον στην αρχική συζήτηση για την επαρκή πρεκοδότηση. Αυτό δεν αποκλείει το να διερευνήσουμε νέες πηγές τις φορές. Αλλά θα πρέπει να δούμε από πού θα αντλήσουμε αυτούς τους πόρους. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο νυφάλιο, με κάποια συμπερασματικά κριτήρια. Επιστρατεύοντας αυτή την ευελιξία για την οποία μιλούμε. Αλλά οπωσδήποτε να πάρουμε χρήματα ούτε από το Connecting Europe Facility ούτε από το Horizon 2020. Ευχαριστώ. Έχει περάσει ήδη η πρώτη ώρα της συνεδρίασή μας. Και ως κοινή προεδρία, επειδή πρέπει να φύγει ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, θα δώσω το λόγο στον Πάμπλο Σάλμπα, που αντικαθιστά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άνεμανς έχει το λόγο, από τους μη γεγραμμένους. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαστε και τόσο ενθουσιασμένοι για αυτό το ταμείο, αλλά υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Πρώτα απ' όλα είναι μια πολιτική απόφαση να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Γι' αυτό υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για τις προτάσεις Juncker. Ο στόχος δηλαδή είναι να υπάρχει αξιόπιστη πολιτική για να έχουμε αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που τόσο το έχουν ε, αναφέρει. Αλλά υπάρχει αβεβαιότητα για το πόση μόχλευση θα έχει. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα και για την ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων τα κριτήρια είναι ασαφή. Λέμε ότι θέλουμε να προσελκύσουμε επενδυτές, αλλά δεν είναι σαφές πώς. Λέγεται ότι θέλουμε καινοτόμε μεθόδους Τίθενται λοιπόν πολλά ερωτήματα, κυρίως για τα επενδυτικά κριτήρια, την επιλογή δηλαδή των προγραμμάτων και την αξιοπιστία τους. Είναι μια και ενσιανή πρωτοβουλία, είναι σαφές αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι η ίδια η φύση της ε, ευρωπαϊκής οικοδόμησης και των δομών. Βλέπουμε τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρωζώνη και αλλού αλλά είναι πολύ πιο έντονα ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης σε σχέση με τα κράτη-μέλη της Ένωσης που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Οπότε, στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις πιέσεις που υφίστανται για να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η ουσία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Άνεμανς. Ο κύριος ε, Κόλμερ, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα να αναφερθώ σε μερικά ουσιώδη στοιχεία. Είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα, συζητάμε για ένα επενδυτικό πρόγραμμα 315 δισεκατομμύρων. Εύκολα λέμε κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε να προωθήσουμε προγράμματα, τι εννοούμε. Θέλουμε να προωθήσουμε προγράμματα το καθένα έχει μέσο, το μέσο μέγεθος των προγραμμάτων είναι 10 εκατομμύρια και τόσο λίγα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να, να χρηματοδοτήσουμε 3.500 προγράμματα. Και αν είναι 1 ε, εκατομμύριο η μέση χρηματοδότηση, τότε θα έχουμε 315.000. Όλα αυτά θα είναι ε, βιώσιμα, θα είναι επικερδή και θα έχουν αποτέλεσμα στην οικονομία. Αλλά εδώ υπάρχουν αντιφάσεις. Όσο καλύτερα θα ακούγεται ένα πρόγραμμα, τόσο λιγότερο θα είναι συμπληρωματικό. Προσθετικό πρόγραμμα δηλαδή, όπως το ορίζει το ΕΦΣΙ. Γιατί αν είναι τόσο καλό, αν είναι τόσο επικερδές, θα το είχα χρηματοδοτήσει και χωρίς το ΕΦΣΙ. Οπότε με πολύ ενδιαφέρον ε, θέλω να δω και πώς θα βρούμε αυτούς τους καταπληκτικούς διαχειριστές οι οποίοι θα μπορέσουν να βρουν, να αποτιμήσουν και να εφαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα 3 έως 30.000 νέα προγράμματα. Δεν μου φαίνεται για τόσο εφικτό αυτό. Ακόμη λιγότερο εφικτό μου φαίνεται, επειδή ακούσαμε και την έννοια έλεγχο. Παρακαλώ, ποιο θα τα ελέγχει όλα αυτά. Ούτε τους κανόνες δεν ξέρουμε. Μπορώ λοιπόν ε, να φανταστώ ήδη τι θα περιέχουν οι εκθέσεις ελέγχου ασαφείς ε, και εφόσον υπάρχει αβεβαιότητα θα είναι όλες οι πολύ θετικές αφού τους δεν ξέρουμε τι να μετρήσουμε. Γι' αυτό, συνάλφε Ούλμαν, θεωρώ πως δεν θα ήταν πολύ καλό να σας δώσουμε τις πιστοτικές μας ε, κάρτες για να υλοποιήσετε τέτοια προγράμματα. Έχω επιφυλάξεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλλη τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές. Γιατί ακριβώ όπω είπε και ο ε, Τζάνι, ε, αυτό αποτελεί βελτίωση του έργου του δηλαδή της πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να δούμε ε, πώ θα αποκρισταλωθεί το θέμα αφού το επεξεργαστούμε. Θέλω να δούμε, υπάρχουν εδώ πέρα κάποια κενά, θα πρέπει να μιλούμε για άλλους ε, πόρου και λέμε για περικοπές στην ε, έρευνα, οπότε θα κατεβάσουμε και τις προτάσεις, γιατί είπαμε ότι θα υπάρξουν διάφορες τέτοιες ε, δαπάνες, αλλά δεν θέλουμε στην καινοτομία και στην έρευνα να έχουν περικοπές. Διαφάνεια όσον αφορά την λήψη των αποφάσεων. Να αποφύγουμε να υπάρχει ένα σύστημα πελατειακό, όπου το δημόσιο χρήμα θα πηγαίνει για το ιδιωτικό όφελος. Άρα θα πρέπει να δούμε για το project financing ποια είναι τα κενά που υπάρχουν γιατί τα έργα και τα προγράμματα τα τελευταία χρόνια τα οποία χρηματοδοτήθηκαν κατέδειξαν ότι υπάρχει στο σύστημα κενό. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα καλυφθεί ο ιδιωτικό τομέα με κάποιο τρόπο να έχουμε εγγυήσει που να καλύπτει. Επίσης ε, για τις ΜΜΕ, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις της καινοτομίας πώς θα έχουμε την ενίσχυσή τους και κάποιους παραπάνω όρους για ούτως ώστε να συμβάλλουμε στην ε, ανάπτυξη. Ε, είπαμε πάλι και δεν αποφύγουμε το πελατειακό σύστημα αλλά να δούμε πώς θα ελκύσουμε κάποιες επενδύσεις για αναθέρμανση της οικονομίας. Και έχουμε 315 δι για τρία χρόνια, δηλαδή περίπου 100 δι τη χρονιά που θα μοιραστούν όλες οι χώρες. Άρα λιγότερο από πέντε δις ανά χώρα. Βλέπουμε μόνο ότι είναι περιορισμένη η επίπτωση. Άρα χρειάζεται κάποιο είδους marketing για να τα διαχειριστούμε και έτσι να αναφερμαθεί επιτέλου η οικονομία. Ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Βάλη, Ο κύριος Ομαρτζή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω τρεις παρατηρήσεις και τρεις ανησυχίες. Η πρώτη μου παρατήρηση και πρώτη ανησυχία αφορά το θέμα της γεωγραφικής κατανομής. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την εθνικοποίηση. Αλλά γιατί να μην έχουμε υπόψη τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Θα ήθελα να καλέσω τις δύο επιτροπές ε, οικονομικών υποθέσεων και προϋπολογισμών να δείξουν κάποια ευαισθησία και στις ε, απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών. Στην γνώμη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών που ήδη έχουν θορυβηθεί γιατί φοβούνται ότι θα γίνει μια συγκέντρωση των πιστώσεων στις μεγάλες Μητροπόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα παραγωνιστούν οι περιφέρειες ε, ε, και οι περιοχές που χρειάζονται περισσότερο τις επενδύσεις. Ας μην ξεχνούμε ότι ο απότερος σκοπός ε, του επενδυτικού σχεδίου του Juncker είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, είναι η ενίσχυση των θέσεων εργασίας. Οπότε θα ήταν παράδοξο να μην επενδύσουμε σε περιφέρειες που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχνούμε τους στόχους της συνοχής στην επιλογή των επενδυτικών σχεδίων. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε και για τη χρήση του θεματικού απόδοσης ή επιδόσεων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το θέμα αφορά την περιφερειακή πολιτική. Γιατί στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία Μιλήσαμε για αυτό το αποθεματικό των επιδόσεων στην Επιτροπή των Περιφερειών και ήμουν παρόν στις διαπραγματεύσεις που ήταν ε, σφοδρές και εξαιρετικά δυσχερείς και πραγματικά δεν θεωρώ ότι μπορούμε έτσι με μια μονοκοντιλιά και χωρίς ε, προφυλάξεις να αναλάβουμε τέτοιου είδους ε, δεσμεύσεις. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και συνετοί. Η δεύτερη μου παρατήρηση αφορά τη διακυβέρνηση. Φυσικά χρειάζεται περισσότερος έλεγχος και μεγαλύτερη διαφάνεια και γι' αυτό θα καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες. Θα μεριμνήσουμε να αποφευθεί και σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ηθινόντων για τη λήψη αποφάσεων και των ιδιωτών επενδυτών. Και τέλος, ένα φλέγο ζήτημα γιατί βρισκόμαστε στην ε, κοινοβουλευτική διαδικασία. Ε, ξεπεράστε το χρόνο σας. Πρέπει να σπεύσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σπεύδει και επιταχύνει τις διαδικασίες, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα συμφωνεί και συνεννοείται με τα κράτη-μέλη, ενώ το δικό μας έργο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και βάρος. Ευχαριστούμε κυρία, κυρία Ομαρτζή. Η κυρία Χιούμπνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούλμαν είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ζήστρο τουρ και λυπάται που τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να συμβάλλουν επίσης στο, στην πολύ χαμηλή κεφαλιακή βάση. Νομίζω ότι αν συνέβαλαν και τα κράτη-μέλη στη βάση εγγύσεων τότε θα υπήρχε θέμα ζήστρο τουρ Οπότε εγώ αν ήμουν επιτροπή θα χαιρόμουν που δεν συμβάλλουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό έχουμε τις επενδυτικές πλατφόρμες όπου μπορούν να συμμετάσχουν. Και επίσης ε, εάν ε, θίξουμε τις εθνικές παρεμβάσεις θα ίσχυε το ζήστρο ετούρ. Οπότε το όλο εγχείρημα θα πήγαινε στράφη. Τώρα, τι είδου έλεγχο προτείνουμε, αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω αν εξέτασα αρκετά προσεκτικά το κείμενο. Αλλά για μένα αυτού του τύπου οι εκθέσεις θα έπρεπε να είναι πιο πολύ εξ άντε στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών για τις επενδύσεις και της στρατηγικής. Έτσι θα ήταν χρήσιμο, γιατί βεβαίως ως αρχή επί του προπολογισμού είμαστε αρμόδιοι για αυτά. Τρίτο σχόλιο, ερώτηση. Οι εγγυήσει που ε, ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστούν, δεν θα μπορούσαν να επανέλθουν στα προγράμματα από όπου έχουν ληφθεί. Και τέταρτον, το είπαν διάφοροι συναδελφοί ήδη, αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των κόμβων συμβούλων. Έχουμε αυτό το Τζάσπερς στην ε, πολιτική συνοχής από το 2007 λειτουργεί σε, σε τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως ε, τέτοιος κόμβος και βλέπουμε ότι η δυνατότητα απορρόφησης και η δυνατότητα προετοιμασίας προγραμμάτων που πρέπει να ανταποκρίνονται σε πολλά περίπλοκα κριτήρια και που θα βασίζονται σε ένα νέο είδος χρηματοδότησης. Βλέπουμε ότι Ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες μας δεν υπάρχει επαρκής τεχνογνωσία. Θα πρέπει πραγματικά να είναι αποτελεσματικός και να βοηθάει ο κόμβος αυτός συμβούλων και όχι να τον αμφισβητούμε ευθύ εξ αρχής. Και τώρα για τις ακροάσεις αυτές στο Κοινοβούλιο. Μα με συγχωρείτε και άλλοι μιλήσαν σχεδόν 4 λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω σοβαρές αμφιβολίες. για αυτές τις ακροάσεις με τους ε, εμπειρογνώμονες. Έχουμε εμπειρία ως έκον. Μα είναι άτομα που θα είναι υπεύθυνα για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Θα είναι τμήμα του συστήματος. Πρέπει λοιπόν την ευθύνη για την επιλογή τους να την δώσουμε ε, σε κάποιο σημείο του συστήματος αλλά όχι Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Μούντι. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ για το εντυπωσιακό έργο των συνεισηγητών και έχουμε και τις ε, τροπολογίες. Τώρα θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της διακυβέρνησης και της υποχρέωσης λογοδοσίας. Και συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους οι οποίοι μας είπαν ότι η φράση εμπιστευτείτε με, είμαι τραπεζίτης, δεν πείθει πια κανέναν. Οπότε γι' αυτό και τόσο το μάλλον είναι σημαντικότερος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση αυτού του κανονισμού και όσον αφορά το πώς μπορούμε να τον αλλάξουμε προς το καλύτερο. η προσθετικότητα και πώς θα καθοριστούν τα, τις διαχείριση είναι πολύ σημαντικά και βέβαια η Επιτροπή των Προπολογισμών αλλά και η Ήτρε θα πρέπει να δουν από πού θα προωθούν αυτοί οι πόροι που αναζητούνται. Και έχουμε την ενίσχυση των, ε, της έρευνας με τις σχετικές υποτροφίες και αυτό είναι πολύ σημαντικό αλλά πολλές φορές Συμβούλιο και Κομισιόν προσπαθούν να παρακάμψουν αυτό το οποίο θέλουμε να ισχύσει αυτήν την χρηματοδότηση αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με τον κόμβο των συμβουλών γιατί αυτό θα πρέπει να εισφέρει κάποια προστιθέμενη αξία όσον αφορά εκείνους οι οποίοι θα αναζητήσουν υποστήριξη από το Ταμείο. Θα πρέπει αυτοί οι ετούντες να έχουν ξεκάθαρα στο μυαλό τους για το τι ισχύει. Επομένως, ε, αυτός ο κόμβος μπορεί όντως να ωφελήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρο, Πρόεδρος, κυρία Μούντι. Ο κύριος κάνει σχετί το λόγο, αλλά δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Οπότε παίρνει το λόγο η κυρία Φερέρα. Δεν θα επαναλάβω τα σχόλια των προλαλισσάντων. Ευχαριστώ και εγώ τους ε, συνεισηγητές. Πολύ αξιόλογο έργο. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε πιο διεξοδικά το κείμενο, γιατί δεν είναι εύκολο να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί όλος ο μηχανισμός. Ε, υπάρχει μια Επιτροπή Επενδύσεων, ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να δούμε τον επιμερισμό των καθηκόντων για να δημιουργήσουμε μια συνολική εικόνα του όλου συστήματος. Επίσης, ε, θα πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα το θέμα της διακυβέρνησης. Γιατί έχουμε το άρθρο 3 αφενός που προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αντανακλά το κεφάλαιο και τις φορές που έχουν κατατεθεί στο Ταμείο και μετά από αυτή την αρχική φάση όπου γίνονται η στρατηγική προσανατολισμή μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε μια μεταγενέστερη φάση πρέπει να μεριμνήσουμε να τηρηθούν αυτοί οι στρατηγικοί προσανατολισμοί και να μην ε, τροποποιηθούν από επενδυτές που θα έρθουν και ε, εκτός από ε, έξωθεν της Ευρώπης ή να ε, μην γίνουν έρμεο της αρχής της δίκαιης ανταπόδοσης. Αυτή η στρατηγική προσανατολισμή. Δεύτερο ζήτημα, τα κριτήρια. Τα κριτήρια κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να περιλαμβάνουν και στόχους για παράδειγμα, τη μείωση των ανισοτήτων, των τεράστιων ανισοτήτων που έχουμε στην Ευρώπη. Γιατί σε μερικέ περιοχέ έχουμε ε, πολλέ επενδύσει ή θα μπορούσαμε να έχουμε, αν το θέλαμε, ενώ σε άλλε περιοχέ, σε άλλε περιφέρειες είναι ανύπαρκτε οι επενδύσει. Οπότε είναι πολύ γενική η στόχη και επίσης έχουμε κάποιες ανεξάρτητες, φορεί ε, φορείς στις και επίσης ένα άλλο εξάρτητο συμβούλιο που θα προβαίνει σε ε, αξιολογήσεις και σε αυτό το ε, συμβούλιο δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Μπορούμε να έχουμε κάποια κρόση και να λαμβάνουμε κάποιες αναφορές, αλλά εκφεύγει του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ε ξεφεύγει του ελέγχου των μελών του Ταμείου των Εγγύσεων. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή πλαισίωση ώστε να μην ξεφύγει ο μηχανισμός αυτός από τους στόχους ε, που επιδιώκουμε. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να δούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα, η συγγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε χαρώ και να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές Φερνάντες ε, και Μπούλμαν για τις εξαιρετικές προτάσεις που περιέλαβα στην έκθεση που είναι και τολμηρές και αποτελεσματικές. Είναι σαφές ότι είναι χρήσιμη η επενδυτική πρωτοβουλία του κ. Γιούγκερ, αυτό είναι αναφίβολο και από τη σκοπιά του τουρισμού και των μεταφορών. Θέλουμε να, να ευοδοθεί αυτό το σχέδιο, το επενδυτικό. Γιατί θα πρέπει να προσανατολιστούμε στις επενδύσεις ε, για ανάπτυξη και απασχόληση. Σημαντικό όμως είναι το θέμα της προσθετικότητας για να μην γδίνουμε κάποιον για να ντύσουμε άλλον. Να μην παίρνουμε από τη μία τσέπη για να τα βάλουμε στην άλλη. Και εκεί είχαμε δύο σημαντικά επενδυτικά ενωσιακά εργαλεία για τη στρατηγική του 2020, το συνδέοντας την Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020 ε, εξαιτία αυτή τη σπουδή τη βιασύνη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει εύκολε λύσει για τη χρηματοδότηση, απορρόφησε κάποια κονδύλια από αυτά τα δύο μέτρα. Ε, Μοιραίο λάθο, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δύο εργαλεία. Θα αποδυναμωθεί τελείω το συνδέοντα στην Ευρώπη, αν αφαιρέσουμε κονδύλια από εκεί. Και επίση ε, θα δώσουμε πολύ συγκεχημένα μηνύματα ε, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα υλοποίηση των στόχων της ε, στρατηγικής του 2020, αποδυναμώνοντας το συνδέοντα στην Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020. Επίσης, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανακτήσει τη λειτουργία του. Δηλαδή, να προσπαθήσει να βρει χρηματοδότηση. Είμαστε εμπειρογνώμονες, ειδικοί στο θέμα αυτό. Το είδαμε ε, και με το πρόβλημα των πληρωμών, ότι μπορούμε να βρούμε με αποτελεσματικό τρόπο χρηματοδότηση. Επίσης, όπω είπε ε, ένα συνάδελφο, δεν έχουμε Ευρωπαϊκό Ταμείο ουσιαστικά στρατηγικών επενδύσεων, αλλά Ευρωπαϊκέ Εγγύσει στρατηγικών επενδύσεων. Οπότε για, για τι εγγύσει μπορούμε να είμαστε πολύ ευρηματικοί. Γιατί φτάσαμε μέχρι τα δύο πρώτα χρόνια, θα πρέπει να δούμε και τι μέλη γενέστε μετά το τρίτο τέταρτο χρόνο. Επίση, το συνδέοντα στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό στο πρώτο ε, διαγωνισμό των σχεδίων. Για τη διακυβέρνηση, σημαντικέ εθνικέ πλατφόρμε για να συγκεντρώσουμε χρήματα και να επιλέξουμε βιώσιμα σχέδια, ενδιαφέροντα και φυσικά σχετικά πολύμορφα. Οπότε και στο Συνδέοντα στην Ευρώπη θα επικεντρωθούμε και στους διαδρόμους αλλά και στις ε, υποδομές, ενισχύοντας σχέδια που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τους ε, εμπειρογνώμονες ε, του χρηματοπιστωτικού κλάδου, δεν θα πρέπει να είναι μόνο εμπειρογνώμονε του χρηματοπιστωτικού κλάδου, αλλά διαφόρων κλάδων. Αναφέρθηκε το θέμα των εισφορών των κρατών μελών. Επίσης, το σύμφωνο σταθερότητα δεν θα πρέπει να γίνει εμπόδιο για την συμμετοχή στην πρωτοβουλία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Γιάλα. Ο κύριος Βιέγας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επισημάνω τις ε, σημαντικές ε, διαφορές και διαφωνίες που έχουμε στην ΚΟΕ για την ουσία του θέματος ε, για τα βασικά χαρακτηριστικά και τους τρόπους χρηματοδότησης. Έχουμε ένα διέξοδο. Έχουμε επενδύσεις γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, δεν, υπάρχουν, δεν, έχουμε, δεν υπάρχει καν εμπιστοσύνη και γι' αυτό θα πρέπει να διαπιστώσουμε με την ερμηνεία αυτή ότι αυτό που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια κεϊσιανή λύση δημόσιων επενδύσεων που θα μπορούσε να ε, μας ε, βγάλει από αυτό το αδιέξοδο το οικονομικό. Αυτό όμως το οικονομικό αδιέξοδο οφείλεται στην έλλειψη προπτικής ε, των οικονομικών φορέων που έχουν συρρυκνωθεί και είναι αναμενόμενο. Εγώ είχα επαφές με πολλούς ε, μικρομεσαίους επιχειρηματίες της ε, Πορτογαλίας. Και αυτή η προοπτική της ε, απόλυτης απελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών και της, του ακρεφνούς, της ακρεφνούς σε παγκόσμιο επίπεδο δεν δημιουργεί κανένα λόγο αισιοδοξία στους επιχειρηματίες. Και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει υποτίθεται μία ε, λύση της αγοράς, ενώ η αγορά είναι δυσλειτουργική, η αγορά έχει αποτελεματωθεί, δεν θεωρώ ότι θα τελεσφορήσει και σίγουρα δεν ε, δημιουργεί προοπτικές. Επίσης δεν καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι τον ίδιο προβληματισμό έχουν ε, οι πολίτες, δεν καταλαβαίνουμε πώς η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα μπορεί να αγοράζει μαζικά ομόλογα κρατικού χρέους και από την άλλη δεν έχει κονδύλια για να χρηματοδοτήσει τις δημόσιες επενδύσεις. Αυτό το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτή είναι ουσιαστική διαφορά που μας χωρίζει με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Αλλά είναι χαρακτηριστική του τρόπου λειτουργίας δυστυχώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η πρόταση. Πολλέ αφιβολίε έχουμε ω προ τη διακυβέρνηση επίση, ω προ τον τρόπο αξιολόγηση ως προς τις ε, εγγυήσει ε, για την ε, ακριβοδίκαιη κατανομή των κονδύλιων. Δεν έχουμε εθνικές ποσοστώσεις. Γιατί? Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το μοναδικό κριτήριο που θα εξασφάλιζε μια ακριβοδίκαιη λύση και θα ενίσχυε την εδαφική συνοχή που τόσο επιθυμούμε όλοι και κοπτόμαστε γι' αυτή. Επίσης, το μοντέλο χρηματοδότησης των υποδομών που στηρίζεται σε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα είναι επίσης ένα μοντέλο που κατά τη γνώμη μας είναι συζητήσιμο. Ευχαριστώ. Ο, η κυρία Άρινα Χίλη. Μίρατζιλ. Ναι, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετώ. Σχετίζω αυτές τις προτάσεις και ευχαριστώ τους συνεισηγητές για το κείμενο τους. Και συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα ήδη είπαν οι συνάδελφοι οπότε και θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, μια που συναποφασίζουν για τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να έχουμε λέγει όσον αφορά την διαχείριση αυτών των έργων και προγραμμάτων. Ακριβώς όπως είπαν οι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να υπάρχει ευελιξία για, για τη χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να εισφέρουν τα κρατημέλια έτσι να ισχυροποιήσουν το Ταμείο. Και όλα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν με ευελιξία όσον αφορά του εθνικού προπολογισμού. Τώρα, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογή, θα πρέπει να καθορίσουμε κάποιε προτεραιότητε που είναι ανάπτυξη και απασχόληση. Όπω είπαν και όλοι οι συνάδελφοι, θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μα στο θέμα το, της ενέργειας, των μεταφορών και εγώ συμπληρώνω την δημιουργική πολιτιστική βιομηχανία το γιατί νομίζω ότι σε αυτό τον τομέα μπορούμε να έχουμε απόδοση και σε ανάπτυξη και σε θέσεις απασχόλησης. Άρα τα κριτήρια μας θα καλύψουν και αυτό τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, κύριε Αγγίλ. Η κυρία Μπάιντερ. Ε, Paldies, priekšsēdētāji. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, Φερνάνδες και Μπούλμαν. Με την έκθεση αυτή γίνεται πολύ πιο σαφής ε, η κατανόηση του όλου εγχειρήματος. Πού θέλω να εστιάσω τώρα. Πρέπει να στηρίξουμε τη συνοχή και χαίρομαι που το αναφέρει η έκθεση οι στόχοι της πολιτικής συνοχής είναι θεμελιώδεις και παίζουν ουσιώδη, θεμελιώδη ρόλο σε πολλές χώρες. Και θα πρέπει ακριβώς ε, στις χώρες με χαμηλότερο ΑΕΠ να χρηματοδοθούν τέτοια προγράμματα για να μην αυξηθεί περαιτέρω το χάσμα. Δεν θα επιτύχουμε τους στόχους ε, της πολιτικής συνοχής μας. Δεν θα ενδυναμώσουμε την οικονομία, δεν θα αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα κτλ οι προηγούμενοι συνάδελφοι είπαν ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι σαφή για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τα σωστά προγράμματα. Συμφωνώ και εγώ. Και επίσης συμφωνώ ότι παρά το ότι θα είναι ανεξάρτητος ο φορέας που θα ελέγχει τα προγράμματα χρειαζόμαστε έναν άλλον μηχανισμό για αποτίμηση της εφαρμογής των προγραμμάτων. Να ενισχυθεί αυτός ο μηχανισμός. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο κόμβος ε, τεχνικών συμβούλων διότι οπωσδήποτε ε, οι χρηματοδοτήσεις για αυτό το νέο πρόγραμμα δεν πρέπει να μειώσουν ε, τις χρηματοδοτήσεις του ε, ε, μέσου συνδέοντας την Ευρώπη διότι χρηματοδοτεί υποδομές που είναι πάρα πολύ σημαντικές δρόμους κτλ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αυτές οι εγγύησεις. Οι εγγυήσεις αυτές είναι ουσιώδεις για να χρηματοδοτήσουμε τέτοια προγράμματα. Επίσης, είμαι υπέρ της ιδέας ότι πρέπει να υποστηριχθούν προγράμματα υψηλότερου κινδύνου. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η Ευρώπη μπορεί να θεωρεί ότι είναι στην πρωτοπορία της καινοτομίας ε, και της επιχειρηματικότητας αλλά δυστυχώς δεν ισχύει πια λόγω ακριβώς αυτής της ε, ε, απροθυμίας να, πάρουμε, να αναλάβουμε κινδύνους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόιρε, συντάκτης γνωμοδότης της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως εισηγητής της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού τη γνωμοδότηση δηλαδή, θέλω να πω ότι για τη χρηματοδότηση να μην ξεχνάμε, όπως ήδη αναφέρθηκε, πόσο δύσκολες ήταν οι συζητήσεις για τις ε, μεσοπρόθεσμες ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Και στην προηγούμενη θητεία και η Επιτροπή Προπολογισμών και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, τότε ήμουν και πρόεδρος της μάλιστα, παλέψαμε μαζί ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να έχει περισσότερη επιρροή. Ότι αυτά που μένουν στη, στον προπολογισμό να είναι αρμοδιότητά μας. Ότι πρέπει οι πιστώσει μα, οι μας να αξιοποιούνται καλύτερα. Και είδαμε ότι κυρίω του τομεί, ε, όπου υπάρχει κοινή αρμοδιότητα, δηλαδή όπου συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη, εκεί κυρίω δεν εκταμιεύονται οι πιστώσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι αποφάσεις για να αφαιρεθούν πόροι από την τεχνολογία και την έρευνα είναι λανθασμένες γιατί σε αυτές τις γραμμές του προπολογισμού η χρήση, η εκταμίευση η αξιοποίηση ήταν καλή. Χρειάζονται λοιπόν αυτοί οι πόροι και στο μέλλον. Δεύτερον, που το προτείνουμε και μέσω τροπολογιών στη γνωμοδότησή μας, είναι το θέμα της εξέτασης, του ελέγχου, της υποχρέωσης λογοδοσίας. Έχουμε δυνατότητα ήδη μέσω του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου να έχουμε εκθέσεις και αποτιμήσεις για τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Τράπεζα Επενδύσεων. Πρέπει να ισχύει και για το ΕΦΣΙ αυτό. Πρέπει δηλαδή να διεκδικήσουμε το ελεκτικό συνέδριο να ελέγχει τα προγράμματα του ΕΦΣΙ για να έχουμε μία εκ των υστέρων αποτίμηση των προγραμμάτων για να μπορεί ακριβώς το Κοινοβούλιο να είναι σίγουρο ότι λογοδοτεί και έναντι των φορολογουμένων για το εάν και κατά πόσο τα προγράμματα αυτά βοήθησαν τους επιδιωκόμενους στόχους. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν οπωσδήποτε ένας φορέας ο οποίος εκ των υστέρων μετά την εφαρμογή να κάνει αποτίμηση της σκοπιμότητας και καλής χρήσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάνικα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την τεράστια προστιθέμενη αξία τους που προσέφεραν στην έκθεση αυτή. Και όλοι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε αυτό το σχέδιο για να μπορέσει να λάβει σάρκα και οστά. Και αν ε, μεταλαμπαδεύσουμε αυτό με τον ενθουσιασμό στην αγορά, τότε η μόχλευση θα ξεπεράσει ακόμη και τα 315 δις που επιθυμούμε. Το επενδυτικό σχέδιο του Juncker είναι ένα, μια ψηφίδα ενός ευρύτερου ψηφιδοτού που θέλουμε να προωθήσουμε. Και στα βήματα που πραγματοποιούμε θα πρέπει να λαμβάνουμε ταυτόχρονα πληροφορίες και για τα άλλα κομμάτια του ψηφιδωτού. Γιατί έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για την Ευρώπη, αλλά οι δράσεις μας ε, θα πρέπει να δούμε τι συνέπειε θα έχουν ακόμη και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Η κυρία Χιούμπνερ κάλεσε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν. Όταν επενδύουν όμω τα κράτη-μέλη και το κατά πόσο θα επενδύσουν θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχημένα θα είναι τα άλλα μέτρα που θα υιοθετήσουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε συνέργειε. Η πατρίδα μου, η μικρή Σλοβακία, ε, θα επωφεληθεί ιδιαίτερα, κυρίως οι 250 επιχειρήσεις που δεν ε, έχουν έδρα σε φορολογικές παραδείσους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Κοραμβάν Χόιζεν, Νόησαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με τα περισσότερα από όσα ακούσαμε από τους συναδέλφους και απλώς θέλω να προσθέσω μια παρατηρησούλα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τον κίνδυνο της ε, ευξημένης πολιτικής παρέμβασης. Τώρα μιλούμε για κάποια προγράμματα και εργαψηλού κινδύνου, οπότε γι' αυτό είπαμε να έχουμε ε, μια επιδυτική επιτροπή, ούτω ώστε τα 3α της αξιολόγησης της ε, ΕΤΕ να μην ε, ανατραπούν. Οπότε θα πρέπει να δούμε πού θα αντλήσουμε πόρους και οπότε θα πρέπει να γίνει επίσης μια σοβαρή συζήτηση για τα σχετικά κριτήρια. Πάντως, μέχρι εκεί. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα χαθεί η των τριών α τη Πενθυγή Τράπεζα. Αυτό θα είναι πολύ κακό. Αυτό ήθελα απλώ, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλει κάποιο συνάδελφο τον ε, λόγο, να τον ζητήσει. Ιδάλω δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Τράπεζα Επενδύσεων και τους συγκητές. Και εδώ και το λόγο κυρίως ε, Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας ε, Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τους συνεισηγητές γιατί εργάστηκαν με ταχύτητα και αυτό δείχνει ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι και για το Κοινοβούλιο θέμα προτεραιότητας. Τώρα θα εστιάσω την προσοχή μου σε εκείνα τα σημεία που είναι περισσότερο προβληματικά. Πρώτα πρώτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός εργασιών όπως ξεκίνησε. Και επίσης να δούμε τι θα γίνει και με ποιες διαδικασίες θα έχουμε τους ορισμούς και διορισμούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ξεφουσκώσει το πράγμα σιγά σιγά. Οπότε όσον αφορά τώρα τις καθημερινές γραμμές για τις ε, επενδύσεις είναι πάρα πολύ θετικό το ότι εσείς ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για αυτή την επενδυτική πολιτική. Αλλά βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι. Άρα για τη συναπόφαση να έχουμε κάποιες καθημερινές γραμμές. Όλες οι κοινωνικές επιτροπές και τα κράτη-μέλη θέλουν να αναλύσουν το θέμα στην ε, κάθε του λεπτομέρεια. Τότε όμως θα χρειαστούμε εξάμεινο, ίσως και χρόνο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση. Οπότε και έτσι θα επιβραδυνθεί πάρα πολύ η εξέλιξη. Και καταλαβαίνω ότι είναι θεμητό αυτό σας το ενδιαφέρον, αλλά παρακαλώ τον παράγοντα ταχύτητα, ρυθμού πρόοδου ούτω ώστε να ολοκληρωθεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε να το έχετε υπόψη. Τώρα όσον αφορά την επιλεξιμότητα, σχετικά κριτήρια επιλογής δηλαδή, νομίζω θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο σε αυτό το σημείο το κείμενο. Ας πούμε εκεί που λέει για κάποια μελέτη επιπτώσεων σε όλη την οικονομία για κάθε έργο και πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή Επενδύσεων. Αυτό είναι κάποιος υπερβολικό. Για Σκεφτείτε. Ε, ας πούμε 25 ανεμόμυλους ή τέλο πάντων έργα αιωλικής ενέργειας σε κάποια χώρα και αυτό να αναλυθεί ε, θα αναλώσει πάρα πολύ χρόνο ή δεν θα ωφέλεις κανέναν τόση ανάλυση. Επίσης, κάτι το οποίο ανέφεραν πολλά μέλη των δύο επιτροπών το πώς θα εξασφαλίσουμε αυτή η επενδυτική επιτροπή να είναι υπεράνω υποψίας. Είναι ακρογωνίας λίθος για αυτή τη ρύθμιση η επιτροπή αυτή και γι' αυτό και θέλουμε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από εμπειρογνώμονες, από κάποιους που να είναι ανεξάρτητοι από την Κεντρική Τράπεζα, την Κομισιόν ή τα κράτη-μέλη και αυτοί να επιλέγονται επί τη βάση των τεχνικών τους γνώσεων. Οπότε και μας προβληματίζει λίγο η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής. Mm. Έτσι νομίζουμε ότι θα πολιτικοποιηθεί η σχετική διαδικασία επιλογής. Εμείς δεν θέλουμε να τους προσλάβουμε για να χαράξουν κάποια πολιτική, κάποιες κατευθυντικές γραμμές. Θα τους επιστατεύσουμε για την υλοποίηση των πολιτικών και των κατευθυντηρίων. Γι' αυτό σας λέω, θέλουμε να εξασφαλιστεί ότι αυτοί θα ενεργούν λαμβάνοντα υπόψη τα του έργου ή του προγράμματος και τίποτα άλλο. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο μείγμα εμπειρογνωμοσύνης για μεταφορές, για ΜΜΕ, για για ενέργεια να υπάρχει επομένω τέτοια πολυμορφία και όλοι μαζί να γνωρίζουν και τα, της γεωγραφίας μια που θα γίνονται σε όλα τα κρατημέλη οι επενδύσεις αλλά όχι, όχι η πολιτική πανέμβαση τελευταίο αλλά σημαντικό τώρα από δική μας πλευράς μας προβληματίζει αρκετά η απάλληψη των άρθρων 18 και 19 ξέρω ότι δεν σας εκπλήσω με τα λόγια μου και να σας τονίσω τα εξής η επιλογή του πώς θα χρηματοδοτηθεί το Ταμείο Εγγύσεων από την αιτήση της για τον προϋπολογισμό θα μας οδηγεί σε μεγαλύτερο από το σημερινό χάος. Ξέρουμε σε την αιτήσια συζήτηση ότι αναζητούνται με τα μεγάλες δυσκολίες τα χρηματοδοτικά περιθώρια. Δεν ξέρω αν το έχετε επισημάνει αυτό, αλλά έτσι δεν θα υπάρχει προβλεψιμότητα για την λειτουργία του ίδιου του προπολογισμού. Μα οι δαπάνες εξαρτώνται από το να μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικό πολιετή προγραμματισμό. Και αυτό κατεξοχήν αφορά την έρευνα. Μα αν δεν ξέρουμε τι θα γίνεται, αν δεν ξέρουμε τι θα περικόψουμε, τι θα γίνει, πώς θα γίνεται η εφαρμογή η υλοποίηση τέλο πάντων των δαπανών. Μα είναι κίνδυνο αυτό. Τώρα κάτι τελευταίο αναφέρετε και εσεί. αυτό που είπατε για την αξιολόγηση της ε, Τράπεζας Επενδύσεων μα θα κινδυνεύσει η αξιολόγηση της ίδια τη Ευρωπαϊκής Ένωση, για να δεν έχουμε κάποιο ξεκάθαρο πλαίσιο που να ρυθμίζει τις σχετικές εγγύησει. Είναι ακαθόδες το θέμα. Δύσκολη η συζήτηση, αλλά δεν μπορούμε να, να κουκουλώσουμε τα προβλήματα και να τα παραπέμψουμε στις καλένδες των ετησίων συζητήσεων του προπολογισμού. Γιατί φυσικά ο καθένας είναι θεμητό να έχει τις απόψεις του πάνω στο τι προτείνουμε εμείς. Όμως, εάν δεν δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, τότε οι αγορές θα μας τιμωρήσουν και ε, το σχέδιό μας θα γνωρίσει δύσκολες ώρες. Όντως κύριε Άντζελ. Τώρα το λόγο έχει εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Uh, uh, ε, λέγομαι Νίκος Τζένετάιμ. Είμαι επικεφαλής του τμήματος ε, για τα νέα προϊόντα στην Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα να πάρω το λόγο. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές, τους ομιλητές για την διαπίστωση που έκαναν ότι οι εγγυήσει που θα δει η Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του ΕΦΣΙ πρέπει να είναι αμετάκλητη και άνευ συνθήκων. Πολλοί ομιλητές το είπαν και εγώ συμφωνώ, είναι θεμελιώδες. Θεμελιωδέστατος. Στόχος των εγγύσεων του ΕΦΣΥ είναι να επιτρέψει στην Τράπεζα Επενδύσεων να αυξήσει τη δυνατότητα να επενδύει σε προγράμματα υψηλότερου κινδύνου και έτσι να μοχλεύσει και τις ιδιωτικές επενδύσεις για να έχουμε αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Για να μπορεί να το κάνει αυτό η ΕΤΕ, ο ρόλος των εγγυήσεων είναι απολύτως θεμελιώδης και οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης που είναι η απόλυτη θεματοφύλακες αυτών των θεμάτων ε, είναι αυστηρή. Άρα οι εγγυήσει πρέπει να είναι αμετάκλητες και άνευ συνθήκων. Ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε. Δεύτερον, η ΕΤΕ αναγνωρίζει πάρα πολύ το ρόλο των εθνικών τραπεζών που θα δώσουν χρηματοδοτήσεις και το ρόλο που θα παίξουν στα πλαίσια του ΕΦΣΥ και θεωρούμε ότι είναι επίσης θεμελιώδης σημασίας η διαχείριση των εγγύσεων όπως προβλέπει και η πρόταση να γίνεται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Τράπεζας Επενδύσεων και να δίδονται έτσι αυτές οι εγγύσεις στις εθνικές τράπεζες προώθησης μέσω διαφόρων πλατφορμών που θα διαχειρίζεται μαζί με τις εθνικές τράπεζες η ΕΤΕ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει συνέπεια στο όλο πρόγραμμα παντού στην Ευρώπη και είναι και η καλύτερη ασφαλιστική δικλίδα κατά των ανησυχιών που πολλά μέλη εξέφρασαν για την ε, ενδεχόμενη επιστροφή της αρχής της δίκαιας επιστροφής, just retour. Ε, βέβαια πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι εθνικοί προωθητικοί τραπεζικοί οργανισμοί σε όλες ε, τις χώρες, άρα είναι θεμελιώδες να μπορεί και από μόνη της η ΕΤΕ να διαχειριστεί αυτές τις εγγύσεις. Τρίτον, Υψηλός κίνδυνος και προσθετικότητα. Όπως πολλοί ομιλητές τόνισαν, ο στόχος του ΕΦΣΥ είναι να μπορεί η ΕΤΕ να διακινδυνεύσει περισσότερο για να επιτευχθεί αυτή η προσθετικότητα και να έχουμε κυρίως ιδιωτικούς επενδυτές. Γι' αυτό λοιπόν να δούμε τα στοιχεία. Τι σημαίνει ακριβώς το εύση. Προσπαθεί να αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό μια σειρά από πρωτοβουλίες που ήδη η τράπεζα έχει επιτυχώς εφαρμόσει σε συνεργασία με την Κομισιόν. Χρησιμοποιώντας ε, ενωσιακούς υπόρους της Επιτροπής ε, με παρόμοιο τρόπο. Πολλά υπόθηκαν για την έρευνα και την καινοτομία και το κενό καινοτομίας να σας υπενθυμίσω το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμά μας που ήδη αξιοποιεί πόρους του ορίζοντα 2020 το Inofin που είναι χρηματοδοτικά μέσα για την έρευνα και την καινοτομία και την ανάπτυξη που βασίζεται σε ένα άλλο πρόγραμμα τη δυνατότητα μέσω του FP7 για τον, την κατανομή κινδύνου. Όλα αυτά είναι οι διαβεβαιώσεις που μπορούμε να σας δώσουμε ότι ε, τα χρηματοδοτικά μέσα που σας προτείνουμε μπορούν να έχουν αποτελέσματα. Και τι σημαίνει προστατικότητα. Προστατικότητα σημαίνει να μπορέσουμε να επεκτείνουμε αυτά τα προγράμματα αναλαμβάνοντας κινδύνους που είναι πέρα από το σύνηθες επίπεδο ε, ανάληψης κινδύνων από την ΕΤΕ αλλά ε, είναι στο επίπεδο ανάληψης κινδύνων που έχουν τα καινοτόμα προγράμματα. Μέσω του ΕΦΣΕ θα μπορούμε να αναλάβουμε τέτοιου κινδύνους. Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στην ανεξαρτησία για τις επενδύσεις αυτές και νομίζω ότι μπορώ, ελπίζω, να σας καθησυχάσω ιδιαίτερα. Κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα επενδύσεων που θα θεωρείται επιλέξιμο μέσω των εγγύσεων ή που θα εγκρίνεται Κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα επενδύσεων λοιπόν θα εγκρίνεται όπως εγκρίνονται όλες οι χρηματοδοτήσεις ε, της ΕΤΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ. Άρα θα έχετε την ε, πλήρη εγγύηση των διαδικασιών της ΕΤΕ για το κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα στο οποίο θα επενδύουμε και το οποίο θα λάβει εγγύσεις μέσω του ΕΦΣΥ. Νομίζω ότι αυτή είναι η απόλυτη εγγύηση ανεξαρτησίας που είναι <coughs> καταχωρημένη στην ε, διακυβέρνηση του ΕΤΕ και από τεχνική και από χρηματοπιστωτική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά πρέπει να σας χορηγεί κάθε διαβεβαίωση που θα θέλατε. Καταλαβαίνουμε τη σημασία της συνοχής. Είναι στόχος κλειδί για το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε πολύ στενά. Στα πλαίσια της συνολικής δανειοδότησής της ε, έχει πολύ αυστηρά κριτήρια λήψης υπόψη της ε, συνοχής τα οποία περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα επενδύσεων. Και τέλος να δώσω το λόγο στους συζητητές μας, πρώτα στον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους ε, για τις προτάσεις τους, ε, να επαναλάβω τις ευχαριστίες ε, και στο προσωπικό στους υπαλλήλους μας, τους βοηθούς, στη γραμματεία για τις εργόδεις προσπάθειες που κατέβαλαν και ε, όπως είπα παρά το πιεστικό χρονοδιάγραμμα έγιναν εκτενείς συζητήσεις γιατί μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το επενδυτικό σχέδιο και γι' αυτό ήταν σημαντικό να προβλέψουμε επαρκή χρόνο για τη συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά και τους και ηγητές για τις, συμβουλές, για τους και τον συνεισηγητή Ούντο Μπούλμαν το συνοδοιπόρο μου σε αυτή την προσπάθεια. Και Ευελπιστώ ότι θα ευοδοθούν οι προσπάθειές μας, γιατί με το Ταμείο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει κερδισμένη και ως προς την ανάπτυξη και ως προς την απασχόληση. Και δεν έχει σχεδόν ε, τίποτα ή ελάχιστα να χάσει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Μόνο 8 δισεκατομμύρια ε, βάζουμε ως εγγύηση για να ε, δημιουργήσουμε μόχλευση και να προσελκύσουμε επενδύσεις ύψους 315 δισεκατομμύριων ευρώ είπαμε στην έκθεση ότι το πλεόνασμα από τα κέρδη του Ταμείου θα επιστρέψει στις γραμμές από τις οποίες προήλθε. Και το θέμα των καταξιδότηση πράξεων είναι ένας τρόπος ε, για να εμπλέξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην όλη διαδικασία. Προβλέπεται καταξιδότηση πράξη για τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνοχή το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, ενισχύει την ε, κοινωνική και την εδαφική συνοχή. Θα καλύψουμε κενά της ε, αγοράς και τα, οι χώρες συνοχής θα έχουν με το Ταμείο αυτό πολύ περισσότερες επενδυτικές δυνατότητες και με το Ταμείο αυτό θα έχουμε προστιθέμενη αξία και με επενδυτικές πλατφόρμες θα επικουρήσουμε και τα διαρθρωτικά ταμεία. Και αυτός ο κόμβος των επενδυτικών συμβουλών είναι πολύ σημαντικός. Και ιδιαίτερα σημαντικός είναι για τις ε, μειονεκτικές περιοχές και για τα κράτη-μέλη της ε, πολιτικής συνοχής. Ο κόμβος αυτός των επενδυτικών συμβουλών θα συμβάλλει στην διάρθρωση προγραμμάτων σε περιφέρειες που δεν έχουν επαρκή διοικητική ικανότητα ή τη δέουσα εμπειρία σε ό,τι αφορά πραγματοποίηση ε, εφαρμογή τέτοιων σχεδίων. Οπότε συνάδει και με την κοινωνική και ταφική συνοχή το ΕΦΣΥ. Μιλήσαμε για τις εγγύσεις, μιλήσαμε για τον προϋπολογισμό. Ε, να ρωτήσει για την διαδικασία επιλογής των ε, προγραμμάτων. Δεν θέλουμε πολιτικοποίηση της διαδικασίας, αλλά ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προσδώσουμε νομιμοποίηση στο ΕΦΣΥ. Σε ό,τι αφορά το τριπλό α, την ε, αξιολόγηση της ΕΤΕΠ, η δική μας πρόταση δεν διαφέρει από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συνδέοντα την Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020 είναι να μειώσει τις αναλήψεις υποχρεώσεων. 2,7 μείωση στο ορίζοντα 2020 και 3,3 δισεκατομμύρια μειώνει από το συνδέοντας την Ευρώπη. Και δίνει και ένα περιθώριο 12 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεν φαίνεται καν στον κανονισμό. Ενώ ο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με, παρά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθεί να βρει μία λύση στην τακτική ετήσια διαδικασία που κινούμε το Συμβούλιο. Εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημάναμε την ανάγκη να έχουμε στην έκθεση και όχι στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ανάγκη να έχουμε μία εγγύηση που θα είναι αμετάκλητη μία ανεγγύηση που θα είναι ανεφόρον. Γιατί θέλουμε το επενδυτικό σχέδιο, λέμε ναι στο επενδυτικό σχέδιο και λέμε ναι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που θέλουμε ήδη να αρχίσει να λειτουργεί από τον Ιούνιο. Οπότε είμαστε υπέρ. Σε ό,τι αφορά το, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σίγουρα μας βοηθά ιδιαίτερα. Γιατί αν αναλάβανε τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ η Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσαμε εμείς να αναλάβουμε τα 5 δισεκατομμύρια και θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια από την ΕΤΕΠ αν γίνει έτσι η κατανομή των εγγυήσεων και θα επέλεγε τα προβλήματά μας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα ήθελα να απευθύνω και μια έκκληση να, οι προτάσεις που θα υποβληθούν να είναι εφικτέ, να είναι ρεαλιστικές. Να μην υποβληθούν προτάσεις που θα αφισβητούν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που θα υποχρεώνουν σε ομοφωνία στο Συμβούλιο, θα ξανανοίγουν το όλο θέμα. Γιατί κάτι τέτοιο θα έδειχνε ότι είμαστε κατά του επενδυτικού σχεδίου και του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ακούστηκαν πολλές επικοδομητικές προτάσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι η καλή επένδυση δεν είναι η δημόσια ή η ιδιωτική. καλή επένδυση είναι αυτή που επιτείνει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεν είναι μόνο οι δημόσιες επενδύσεις ε, ε, αγαθές, δεν είναι αμαρτία οι ιδιωτικές επενδύσεις. Η καλή επένδυση κρίνεται από τα αποτελέσματά της στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Εμείς θέλουμε εφικτά, βιώσιμα, σχέδια, αποτελεσματικά, που να μπορούν να δρομολογηθούν και να αποφέρουν καρπούς. Επίση, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, εκτό ότι προωθεί τι επενδύσει και στηρίζει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, θα μειώσει τη γραφειοκρατία, θα μειώσει ε, τα εμπόδια τη εσωτερική αγορά. Και αυτό θα κάνουν οι επενδυτικέ πλατφόρμες για την Ενεργειακή Ένωση και για τι διασυνδέσει τη μεταφορέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τελευταίο ο συγητή τη Επιτροπή Προπολογισμών, ο κύριο Μπούλμαν. Ευχαριστώ πολύ. 26 συνάδελφοι πήραν το λόγο, τους μέτρησα και τους ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τον κάθε συνάδελφο για τις επικοδομητικές προτάσεις. Νομίζω ότι θα δω και πώ θα περιληφθούν ε, στις τροπολογίες που ενδεχόμενα θα υποβάλλετε. Τώρα έχω 2-3 λεπτά για να αντιμετωπίσω 26 τοποθετήσει. εν πάση περιπτώσει. Καταρχάς, να στραφώ προς την Κομισιόν και την ΕΤΕ πρώτα απ' όλα και συγχωρήστε με γι' αυτό γιατί πρέπει να αναπτύξουμε μια σωστή σχέση εργασίας και κατανόηση για το θέμα αυτό τις επόμενε εβδομάδες. Κοιτάξτε, αν ε, κάνουμε αυτό που προτείνεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόεδρο πλέον για την επόμενη συνεδρίαση. Ο πρώτος έφυγε πριν ε, χρειαστεί να μου δώσει το πορτοφόλι του. Οι άλλοι δύο θα φύγουν γιατί δεν θα μπορούν να εμπιστευτούν αρκετά το πρόγραμμα. Εάν δεν κάνουμε εμείς πρώτα απ' όλα τα δικά μας τα καθήκοντα, δεν συμβάλλουμε επαρκώς δεν θα υπάρξει αρκετή εμπιστοσύνη. Κάτι για την ε, χρονική συνέχεια. Αν κατάλαβα καλά, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και της ε, Τράπεζας Επενδύσεων είχαν ένα εξάμεινο για να διατυπώσουν τις προτάσεις τους. Ο συνάδελφός μου Ζωζέ Μανέλ και εγώ είχαμε τρεις εβδομάδες για να υποβάλουμε το σχέδιο έκθεσης. Και οι διαρμηνείς μας εργάστηκαν ταχύτατα για να μεταφράσουν τα κείμενα. Σας υπόσχομαι τα εξής δύο. Πρώτον, θα εργαστούμε όσο γρήγορα και όσο αποτελεσματικά μπορούμε μέχρι το όριο της αντοχής των συνεργατών μας και του εαυτού μας. Και σας υπόσχομαι επίσης το εξής, μια για πάντα να το ξέρετε, ότι δεν είναι δυνατόν το σώμα μας να κλείνει τα μάτια και να αφήνει να περνάει ό,τι θέλετε εσείς. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου και αυτό ακριβώς θα κάνουμε που πρέπει. Θα συζητήσουμε μέχρι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τίποτα άλλο δεν θα μπορούσαν να δεχθούν οι ψηφοφόροι μας. Και να διευκρινίσω μια παρανόηση. Σε κανένα κείμενο, σε κανένα στοιχείο του κειμένου που σας υποβάλαμε ο Ζωζέ Μανουέλ και εγώ δεν λέμε ότι το κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα θα πρέπει να εξετάζεται με τόση λεπτομέρεια μέχρι που να έχουν λήξει όλες ε, οι προθεσμίες και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και η ΕΤΕ εξετάζει τα προγράμματα. Θέλουμε όμως να πούμε στην ΕΤΕ να λαμβάνει υπόψη τη συνολική οικονομική επίπτωση του κάθε προγράμματος. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω περαιτέρω. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να τα συζητήσουμε ούτως ώστε να είναι ικανοποιημένη η Κομισιόν με τις διατυπώσεις μας. Μία δεύτερη παρανόηση. Πουθενά δεν γράψαμε ότι το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει για την επιλογή των ε, εμπειρογνωμόνων. Το αντίθετο ακριβώς. Το αντίθετο. Το Κοινοβούλιο παρακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να του υποβάλει ένα κατάλογο τον οποίο εμείς ενδεχομένω να περικόψουμε. Θα σας πούμε δηλαδή, κοιτάξτε, από τις προτάσεις που μας κάνατε, αυτές θεωρούμε ότι είναι οι καλύτερες. Τίποτα περισσότερο. Δεν είναι πολιτικοποίηση αυτό. Επαναλαμβάνω, ο ενωσιακός προϋπολογισμός είναι ο μόνος εγγυητής των αναλαμβανωμένων κινδύνων. Οπότε ο νομοθέτης πρέπει να σκεφτεί να έχει γνώμη και για το ποια άτομα θα διαχειρίζονται τον προπολογισμό. Δεν είναι αυτό καμία παράλογη απέτηση, καμία πολιτικοποίηση. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό καθήκον μία εκπροσώπηση των ψηφοφόρων. Θα έχουμε ευκαιρίες να το συζητήσουμε και περαιτέρω. Υπάρχουν ε, πιο ε, ειδήμονες από μένα για τη μορφή των χρηματοδοτήσεων. Ο Ζωζέ Μανέλ ξέρει περισσότερα και είμαι σίγουρος ότι μαζί θα βρούμε λύση που θα λαμβάνει υπόψη και την ευελιξία, θα λαμβάνει υπόψη και το επίπεδο γνώσης των μελών μας και οπωσδήποτε θα τηρεί και την προϋπόθεση ότι πρέπει το νέο ταμείο να λειτουργεί διαφανώς και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπούλμαν. Έχουμε επίγνωση των ε, ευθυνών του Κοινοβουλίου, γιατί έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλέ προσδοκίε για αυτή την σημαντική υπόθεση. Οπότε δεν υπάρχει χώρος για αποτυχία, δεν πάμε περιθώρια τέτοια. Οπότε θα πρέπει όλοι βέβαια να είμαστε ευέλικτοι για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία η οποία να είναι πάνω απ' όλα υπέρ των συμφωνών των ε, Ευρωπαίων. στον συμπρόεδρό μου τον λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, έχει εντυπωσιάσει η συζήτησή μας. Υπόσχεται πολλά και καταδεικνύει πόσο το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να ανταποκριθεί εντάχει όσον αφορά αυτές τις προσδοκίες των επενδύσεων τόσο ώστε να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε γιατί έχουμε τις εξής προκλήσεις. Πρώτα πρώτα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής της ιδέας γιατί μας επικρίνουν ότι η λήψη των αποφάσεων που ε, γίνεται μετά από πάρα πολύ μακρόχρονες διαδικασίες και ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε όσο γρήγορα επιβάλλει η συγκυρία και πώς δοκούν οι συμπολίτες μας. Όμως ευχαριστώ τους συνεισηγητές γιατί απέδειξαν ότι μπορούμε να κινητοποιηθούμε, να δουλέψουμε γρήγορα, να διατυπώσουμε προτάσεις. Αυτό είναι ελπιδοφόρο για το μέλλον. Δεύτερη πρόκληση να μην έχουμε πολυνομία γιατί έχουμε κάτι σαν κυβέρνηση με κανόνες, με νόμους λειτουργούμε. Όμως θα πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε υπόψη τους στόχους που να πετύχουμε. Και τρίτον είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Άλλη, τρίτη πρόκληση. Έχουμε έλλειψη επενδύσεων αλλά υπάρχει και πολύ ρευστότητα. Οπότε έχουμε τώρα αυτή την ποσοτική χαλάρωση της ε, κοινωνικής Τράπεζας όπου έχει φέρει για τους επενδυτές ρευστότητα μεγάλη δηλαδή δεν έχουν να κάνουν τα χρήματά τους. Οπότε και τι κάνουν με αρνητικά επιτόκια δανείζουν στα κράτη-μέλη. Επομένω, δεν είναι πρόβλημα ε, ρευστότητας αλλά είναι πρόβλημα επιτοκίων. Μιλάμε όμως τώρα για κάποιους είδους κινδύνους που περικλίνουν αυτέ οι επενδύσεις. Άρα θα πρέπει για να πείσουν τους επενδυτές να θεσπίσουν αυτό το Ταμείο Εγγύησης στο οποίο συμπληρωματικά θα μετέχει η ΕΤΕ. Οπότε ε, μου ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η πρόταση των συζητών θα πρέπει τα κρατημέλη κάθε χρόνο δημοσιονομικά να καλύπτουν ό,τι χρειάζεται. Ναι, συναδελφοί, θα αρέσει αυτό στις ε, αγορές. Και θυμάμαι τις τελευταίες διαπραγματεύσεις για τον διορθωτικό προπολογισμό της χρήσης του 14 και το σχέδιο προπολογισμού για τη χρήση 15 και τα καταφέραμε παρά τα 4.800 των επιπλέον πληρωμών γιατί καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε ε, τα μη καταβληθέντα, τα 25 δις. Κάτι το οποίο μπορεί να προβληματίσει τους ε, επενδυτές. Μα αν δεν μπορούν να πληρώσουν αυτά τα 25 δις για αυτά που δεν έχουν πληρώσει στις, στις ταχθείς της μα τι εγγύσεις να δώσουν εγώ. Πιστεύω ότι οι συνεισηγητές θα βρουν κάποια λύση ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια εμπιστοσύνη χωρίς ερωτηματικά. Και η διαγραφή των άρθρων 18 και 19 επιδέχεται διαπραγματεύσεις τις επόμενες εβδομάδες. Αγαπητοί συνάδελφοι, Μπούλμαν και Φερνάνδες. Και οι συγητέ των άλλων επιτροπών, τη Ήτρε και τη Τραν και αυτοί θα βρουν κάποια λύση προβλέψιμη ε, σαφή γιατί μιλούμε για μακρόπνοες επενδύσεις και σε αυτή την περίπτωση οι επενδυτές θέλουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και θέλουν ένα ενιαίο σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτά και πάλι σας ευχαριστώ και πάλι μπράβο σας. Ευχαριστούμε και τους ε, συνεργάτες των ε, δύο επιτροπών μας αλλά και των άλλων επιτροπών γιατί μιλούμε για περισσότερες επιτροπές τώρα που συνεργάζονται οπότε και το Κοινοβούλιο θα καταλήξει σε αυτή την ενιαία πρόταση. Και ελπίζουμε να πείσουμε και το Συμβούλιο να συμφωνήσει. Τροπολογίες. Μέχρι την 5η 19 Μαρτίου το μεσημέρι. Και δεν θα έχουμε χωριστές τροπολογίες σύμφωνα με το άρθρο 59 όσον αφορά το αταφκαπα 4 γιατί προβλέπει ο κανονισμός ότι οι τροπολογίες θα αφορούν την σύμφωνη γνώμη ή την απόρριψη επί της προτάσεως της Επιτροπής. Και θα περιέχουν απλώς πολιτικά σχόλια και όχι άλλου είδους προτάσεις. Σας ευχαριστώ.